Euh, Συνάδελφοι, να συνεχίσουμε τις εργασίες μας στο πλαίσιο της εξέτασης της έκθεσης ε, Τσάμπα Ορή τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησεις των κρατών μελών προβλέψαμε σήμερα χρόνο για την ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Μπρουνό Κοκέ που είναι πρόεδρος της ΕΜΚΟ της Employment Committee στα ωραία γαλλικά μας, στην Επιτροπή Απασχόλησης, το όργανο που από την πλευρά του Συμβουλίου προετοιμάζει τις αποφάσεις της ΕΠΣΚΟ, του Συμβουλίου για τις Κοινωνικές Υποθέσεις. Και η οποία, μάλλον το οποίο, έχει καθοριστική θέση για τις τροπολογίες έτσι όπως αποφασίζονται και περατώνονται από το Συμβούλιο στην εξετάσή του. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που ήρθατε σήμερα να μιλήσετε μαζί μα. και όσοι ήθιστε στα ζώα μα, θα σας δώσω το λόγο για ένα δεκάλεπτο για να μας παρουσιάσετε τη διάθεση και την στάση του Συμβουλίου. Να, μας, να ενημερώσετε μάλλον τα μέλη της Επιτροπής μας και για το χρονοδιάγραμμα, διότι δεν υπάρχει ικανοποίηση από την πλευρά των ε, βουλευτών μας, του Κοινοβουλίου, ως προς την υιοθέτηση των καθευθυντηρίων γραμμών φέτος, ακόμη και αν είναι το πρώτο βήμα πραγματικής υλοποίησης της στρατηγικής του 2020. Μια δέσμευση λοιπόν που δεν φαίνεται όμως να οδεύει ομαλά σε σχέση με τις πολιτικές μας ανταλλαγές. Και ακόμη και αν σε αυτό το κοινοβούλιο έχουμε αγωνιστεί σκληρά ώστε οι κατευθυντήριε γραμμές και οι πολιτικές απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων να θεωρηθούν ένα ενιαίο έγγραφο ως οι κατεξοχήν ε, ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές, τελικά οι αρμοδιότητες της Επιτροπής μας, ε, ε, αυτό συμβαίνει και στο Συμβούλιο, καταλήγουν να διαχωρίζονται στην εξέτασή τους μεταξύ διαφόρων οργάνων. Παραδόξως λοιπόν η Επιτροπή μας φέτος αποφάσισε να μην συντάξει ψήφισμα για τους γενικούς προσανατολισμούς των κοινωνικών ε, πολιτικών και απασχόλησης και τουλάχιστον θέλουμε να περάσουν κάποια συγκεκριμένα μηνύματα ώστε η δυναμική σχέση μεταξύ των κατευθυντηρίων γραμμών, των διαφόρων κατευθυντηρίων γραμμών να είναι η σωστή. Αυτά στο γενικότερο πλαίσιο της στρατηγικής 2020 και με βάση του στόχου για την μείωση της φτώχειας, κάτι που προφανώς απασχολεί πάρα πολύ και τη δική σας την Επιτροπή και βεβαίως προκαλεί το ενδιαφέρον και των μελών της Επιτροπής μας, οι οποίοι τον περασμένο μήνα τοποθετήθηκαν με μια, ένα ψήφισμα που εγκρίθηκε τον Απρίλιο, καθότι είμαστε πεπισμένοι για τη σημασία του στόχου αυτού και την ανάγκη να τον διατηρήσουμε ως ένα στόχο που θα συζητιέται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η εμβέλειά του είναι σημαντική. Σας δίνω λοιπόν το λόγο για ένα δεκάλεπτο και μετά θα περάσουμε στις ερωταπαντήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που προσκαλέσατε την ΕΜΚΟ να παρουσιάσει τις απόψεις σας και τα αποτελέσματα των συζητήσεων για αυτή τη νέα στρατηγική και τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση που πρόκειται να παρουσιαστούν στο Συμβούλιο. Καταρχάς, όσον αφορά τις ανησυχίες σας για το χρονοδιάγραμμα, πρέπει να πω ότι από πλευρά ΣΕΜΚΟ το θέμα του χρονοδιαγράμματος αποτελεί επίσης πρόβλημα. Καταρχάς γιατί καθυστέρησε πολύ η στρατηγική, η πρόταση της Κομισιόν δηλαδή που ήρθε αρχές Μαρτίου, ενώ λίγη η παλαιά στρατηγική στο τέλος του έτους, άρα πρέπει να ληφθεί απόφαση πριν το Συμβούλιο του Ιουνίου. Λάβαμε όμως ε, την πρόταση μόλις πριν ε, το Συμβούλιο το ΕΑΡΙΝΟ και από τη στιγμή που το Εαρινό Συμβούλιο αποφάσισε κάποια πράγματα, η σύνθεση των κατευθυντήριων γραμμών επί των οποίων ε, εργαζόμαστε σήμερα παρουσιάστηκε πολύ καθυστερημένα. Επομένως, στην ΕΜΚΟ συζητήσαμε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές μόνο μία φορά τελικά. Την προπροηγούμενη εβδομάδα. Να πω ότι συζητήσαμε τις κατευθυντήριες γραμμές για μία ολόκληρη ημέρα. Είχε γίνει βέβαια και κάποια προπαρασκευαστική εργασία στις υποομάδες της ΕΜΚΟ, αλλά στην ΕΜΚΑΦΚΑ τι καθεαυτή τη συζητήσαμε μόνο μία μέρα. Σε αντίθεση με αυτό που είχε γίνει για το 2007. Οπότε εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε υπό τις συνθήκες για να καταλήξουμε σε ένα συνενετικό κείμενο. Όμως αυτό έχει κάποιες συνέπειες. Καταρχάς κάτι που έχει να κάνει με τη διάγνωση ότι απέτυχε η προηγούμενη στρατηγική. Αυτή η αποτυχία οφείλεται σε δύο θέματα. Από τη μία πλευρά στο ότι δεν υπήρξε αίσθημα ιδιοκτησίας, αν θέλετε, της στρατηγικής και δεύτερον θέματα που είχαν να κάνουν με την διαχείριση διακυβέρνηση. Το νέο χρονοδιάγραμμα μας επιτρέπει να πούμε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη υιοθέτηση της στρατηγικής. Τώρα, πολλά πράγματα, πολλές πρωτοβουλίες δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή πώς θα υλοποιηθούν, οπότε αυτή τη στιγμή συζητάμε λίγο αφηρημένα τις κατευθυντήριες γραμμές και προσπαθούμε να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται για την ΕΜΚΟ αυτό τα δύο πράγματα σήμαιναν ότι κατά κάποιο τρόπο υπήρξε μία φορτισμένη αν θέλετε ατμόσφαιρα και η συνάντησή μας στην ΕΜΚΟ ήταν περισσότερο αστυνόμευση παρά συζήτηση επί της ουσίας Αυτά λοιπόν όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα και τις πολύ συγκεκριμένες συνέπειές του στην στρατηγική και στο πώς και με ποια εργαλεία θα υλοποιηθεί. Πάντως, είχαμε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, κάτι πολύ σημαντικό για την Επιτροπή Απασχόλησης. Είναι πολύ σημαντικό, καθώς ε, και στην προηγούμενη στρατηγική είχαμε συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. Και βεβαίως, εφόσον αυτός είναι και ο τομέας της Επιτροπής μας, είναι σημαντικό να λάβουμε και τη δική τους άποψη. Τρία πράγματα ελήφθησαν υπόψη στις τροποποιήσεις που έγιναν στη στρατηγική από την Επιτροπή Απασχόλησης στην ΕΜΚΟ. Καταρχάς, οι κοινωνικοί εταίροι ζήτησαν η στρατηγική να μην αφορά μόνο την προσφορά εργασίας αλλά και τη ζήτηση εργασίας, δηλαδή τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης από τις επιχειρήσεις και την ύπαρξη εργαλείων για την εφαρμογή κατάλληλης πολιτικής. Και το δεύτερο θέμα ήταν η μισθή. Είχαν την εντύπωση ότι η διατύπωση που είχε ζητήσει η Κομισιόν ήταν οπισθοδρόμηση σε σχέση με το παρελθόν και η κοινωνικοί εταίροι ήθελαν την αυτονομία τους για τις ε, διαπραγματεύσεις της μισθολογικές. Το άλλο θέμα αφορούσε την ευελιξία. Βεβαίως έχουμε και την κρίση, οπότε ασχοληθήκαμε με τους μηχανισμούς ε, επιδομάτων ανεργίας ε, και άλλων ε, και της μερικής απασχόλησης και όλα αυτά ζήτησαν να ενσωματωθούν περισσότερο με περισσότερες αναφορές στις συνθήκες εργασίας κτλ. Άρα, λάβαμε υπόψη τα αιτήματα των κοινωνικών εταίρων. Περνάω τώρα στις κατευθυντήριες γραμμές αυτές καθ' αυτές. Όπως αναφέρεται στη γνωμοδότηση που εστάλει στην ΕΠΣΚΟ πρόκειται για έναν μακροπρόθεσμο στόχο εδώ που θα μας επιτρέψει όμως να διαμορφώσουμε και την βραχυπρόθεσμη πολιτική μας. Όμως, ο βασικός στόχος της ΕΠΣΚΟ είναι η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης έτσι ώστε το ποσοστό απασχόλησης να φτάσει στο 75% για το ημερίδα του πληθυσμού μεταξύ 25 και 64 ετών του ενεργού πληθυσμού δηλαδή. Επίσης όσον αφορά θέματα όπως την κατάρτιση, εκπαίδευση, αντιμετώπιση της ε, φτώχειας, σε σχέση με την ε, δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Θέλουμε λοιπόν εργαλεία για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης ε, που έχουν ε, εξαφανιστεί ορισμένες φορές. Χρειάζονται λοιπόν οικονομικά κίνητρα και όπως ανέφεραν και οι κοινωνικοί εταίροι υπάρχουν και θέματα που έχουν να κάνουν με τις μισθοδολογικές διαπραγματεύσεις. Άρα, έχουμε τα βασικά. Δημιουργία θέσεων απασχόλησης και επαναφορά στις κατευθυντήριες γραμμές πρωτοβουλίες που θα αναφέρω που έχουν οικονομικές συνέπειες αλλά επιτρέπουν τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Κάτι ακόμη που ανέφεραν οι κοινωνικοί εταίροι αλλά που πιστεύω ότι βρήκε σύμφωνα και πολλά κράτη-μέλη στην ΕΜΚΟ ήταν να είμαστε πιο συγκεκριμένοι στο θέμα της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, στη ζήτηση εργασίας δηλαδή πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με εταιρικέ σχέσεις αλλά όχι μόνο. έβρεση εργαλείων που θα επιτρέψουν την δημιουργία θέσεων απασχόλησης Τρίτος βασικός άξονας που απασχόλησε τα κράτη-μέλη και που ευθυγραμμίζεται με αυτά που ζήτησε η ΕΠΣΚΟ είναι η ισότητα ανδρών γυναικών και η ενσωμάτωσή της πιο συστηματικά και με πιο ευρύ τρόπο. Αναφέρεται στις κατευθυντηρίες γραμμές. Και τονίζεται αυτό το θέμα. Και επίσης ε, η επανασωμάτωση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την ποιότητα της εργασίας, τα κοινωνικά θέματα και την αντιμετώπιση της φτώχειας. Με επανενσωμάτωση των ατόμων στην αγορά εργασίας προκειμένου να επιτρέψουμε τη μείωση της φτώχειας. Αν και αυτό δεν σημαίνει υψηλότερο επίπεδο απασχόλησης υποχρεωτικά, στην ΕΜΚΟ θεωρήσαμε ότι πρέπει να έχουμε ως βάση μία, ένα υψηλό επίπεδο κοινωνικής προστασίας. Άρα, ειδικά η κατευθυντήρια γραμμή 10 δεν θα έπρεπε να αφορά αποκλειστικά την αντιμετώπιση της φτώχειας, αλλά και την αντιμετώπιση της φτώχειας μέσω της ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας των ατόμων που μέχρι στιγμής έχουν αποκλειστεί από αυτήν. Τι άλλο έχει αλλάξει στις κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά το χρόνο. Στην κατευθυντήρια γραμμή 7 έχουμε την ουσία των συζητήσεών μας. Γιατί επειδή αντικατοπτρίζει τι προτείνουμε σήμερα σε σχέση με τη στρατηγική της Λισαβόνας. Η στρατηγική της Λισαβόνας έχει κατευθυντήριες γραμμές ε, για την ε, κατάρτιση, την επαγγελματική κατάρτιση. Και αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές αφορούσαν περισσότερο την εκπαίδευση και την αγορά εργασίας. Τώρα όμως έχουμε περισσότερα πράγματα. Από την άλλη πλευρά όμως έχουμε μείωση στις πέντε κατευθυντήριες γραμμής για την απασχόληση που πλέον έγιναν μία κατευθυντήρια γραμμή για την απασχόληση. Χρειάστηκε λοιπόν να γίνουν επιλογές θέματα όπως η flexicurity, ευελιξία και ασφάλεια αναφέρονται πολύ περισσότερο στις νέες κατευθυντήριες γραμμές. Υπήρξαν λοιπόν πολλές συζητήσεις για αυτή την κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση και υπήρχαν ανησυχίες από τα κράτη-μέλη να μην διαγράψουμε πολλά σε σχέση με το παρελθόν και ότι θα μας επιτρέπουν οι κατευθυντήριες γραμμές να κάνουμε τουλάχιστον αυτά που μπορούσαμε να κάνουμε και στο παρελθόν. Τουλάχιστον αυτά πλούτησαν σε μεγάλο βαθμό όλες τις αναφορές που, χρησιμοποιήθηκαν στις κατευθυντήριες γραμμές. Περισσότερη απασχόληση, περισσότερη δραστηριοποίηση, περισσότερη κινητοποίηση προς την αναζήτηση εργασίας και ε, να μεριμνήσουμε για μισθούς οι οποίοι να δίνουν και κίνητρα και να παρακολουθούν την παραγωγικότητα. Επίσης, πολιτικές δραστήριες για την αγορά εργασίας, για τους ανέργους, για τους νέους χωρίς εργασία. Σε ό,τι αφορά τώρα τις κατευθυντήριες γραμμές για την διαβίου μάθηση και την εκπαίδευση, στις αναφορές μας δεχτήκαμε γενικά τις προτάσεις που μας ήρθαν από την Επιτροπή για την Εκπαίδευση, απλώς φροντίσαμε να ενσωματώσουμε με καλύτερο τρόπο και την μέρημνα για την ενσωμάτωση στον αγορά εργασία, την έναρξη σταδιοδρομία και τη συνέχεια τη σταδιοδρομία των μισθωτών. Άλλο σημείο στη συζήτηση. Που είναι εξόχως σημαντικό ήταν η κατευθυντήρια γραμμή υπαριθμών 10 η γραμμή αυτή, η κατευθυντήρια γραμμή, αποτελούσε πράγματι μια απάντηση στην ε, κοινωνική ρήτρα που εμπεριέχεται στη συνθήκη της Λισαβόνας, σε ό,τι αφορά όμως τη νομική βάση, που η νομική μας βάση αναφέρεται στα θέματα της απασχόλησης, επομένως τα ζητήματα κοινωνικής ενσωμάτωσης θα έπρεπε να κατευθυνθούν προς την ενσωμάτωση των ατόμων στο χώρο εργασίας. Επομένως, η διατύπωση που έχει γίνει ξεκινά με προκατακτικές μνήες που θέτουν στην καρδιά και σαν τελικό στόχο την απασχόληση για την κοινωνική ενσωμάτωση και την ανάπτυξη της κοινωνικής προστασίας και εν γέννη η διατύπωση αυτή έχει σαν στόχο να αποκλείσει διατυπώσεις σε επίπεδο πολιτικής που θεωρούμε ότι δεν συνδέονται με την πολιτική απασχόλησης. Εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει αυτές που δεν συσχετίζονται άμεσα με τον στόχο της επίτευξης της ε, πλήρους απασχόλησης και επίσης η διατύπωση αυτή στοχεύει στο να εξασφαλίσει ότι αυτά που είχαν επιτευχθεί στο παρελθόν με την ενεργοποίηση αυτών των μηχανισμών που ήταν ε, παροτρυντικά στοιχεία για την απασχόληση να μπορέσουν να διατηρηθούν στις νέες κατευθυντήριες γραμμές. Αυτά λοιπόν έχουμε συμφωνήσει για μια πλήρη διατύπωση στα πλαίσια των κατευθυντηριών αυτών γραμμών, αφήνοντας όμως για να συζητηθεί στα πλαίσια του Συμβουλίου το θέμα της στοχοθεσίας, του καθορισμού των στόχων, για την κατάρτιση και την εκπαίδευση και την καταπολέμηση της ε, του κοινωνικού αποκλεισμού και της ένδυας, θέματα που δεν είχαν αντιμετωπιστεί από το Συμβούλιο το, την Άνοιξη, στο Ερενό Συμβούλιο. Είναι τα μόνα στοιχεία λοιπόν τα οποία δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο συμφωνία στην Επιτροπή Απασχόλησης. Αυτά λοιπόν θα μπορούσα να σας πω καταρχήν και φυσικά είμαι διαθέσιμος να απαντήσω στα ερωτήματά σας εάν θέλουν υπάρξει. Σας ευχαριστώ πολύ λέγει η Πρόεδρος. Θα δώσω τώρα το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Τζάμπα Ορί και μετά στην κυρία Στάινεκ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να συνοψίσω εντάχει αυτά τα οποία θέλω να πω και θα πω, κάνω και μερικά σχόλια εν τέλει. Εγώ εξακολουθώ να κατανοώ το ότι το Συμβούλιο καθώς και το Κοινοβούλιο κινούνται σε διαφορετικές τροχές. Το Συμβούλιο έχει καθορίσει το δικό του χρονοδιάγραμμα και τη δική του ημερησία διάταξη και δεν θέλει να αλλάξει πορεία επειδή το Κοινοβούλιο ασχολείται με κάποια άλλα ζητήματα. Προφανώς έχετε δει πρώτα, την πρώτη ε, δομή, της, την πρώτη μορφή ε, του εγγράφου του Συμβουλίου που αποκλίνει από αυτά του, του Κοινοβουλίου μου που αποκλίνει από αυτά που συζήτησε το Συμβούλιο και αυτά που είχε προτείνει η Κομισιόν. Η δική μου άποψη είναι ότι εμείς πρέπει να αναλύσουμε και τις αποτυχίες της ε, ατζέντα της Λισαβόνας και φυσικά μπορούμε να συμφωνήσουμε με αυτά που είπε ο κ. Κοκέτ ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να αντλήσουμε κάποια διδάγματα από αυτή την αποτυχία. Ένα από τα κύρια σφάλματα όμως αυτής της διαδικασίας ήταν το γεγονός ότι οι στόχοι και οι κατευθυντήρε γραμμές για του στόχου του Λισαβόνα είχαν διατυπωθεί με τόσο γενικόλογο τρόπο που να μην υπάρχει κανένα τρόπο παρακολούθηση τη επιτυχία ή όχι σε αυτού του στόχου. Εγώ διάβασα τι εκθέσει των κρατών μελών, όπου το κάθε κράτο μέλο εκπληρούσε συνέχεια όλε τι ε, απαιτήσει. Και όμω, αν συγκρίνουμε τα τελικά αποτελέσματα με αυτά τα οποία είχαμε προβλέψει, πρέπει να δεχτούμε ότι παρασάγκα απέχουν από αυτό το οποίο είχε προβλεφθεί. Αυτό είναι λοιπόν το σημείο κίνησή μου. Εγώ είμαι έτοιμος να χαιρετήσω την ε, παρουσία ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών με κύριο στόχο την βελτίωση της απασχόλησης. Αυτό φυσικά είναι το βασικό μας πρόβλημα και κανείς δεν το αμφισβητεί. Δεν νομίζω ότι ο στόχος 75% συμμετοχή στην αγορά εργασίας είναι υπερβολικός, ακόμα και αν η εφαρμογή αυτού του στόχου προσκρούσει σε κάποιες δυσκολίες. Επίσης δεν είναι οι πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών αυτές καθεαυτές, αλλά η ίδια η οικονομία η οποία θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης. Ο πρώτος στόχος λοιπόν θα πρέπει να είναι η δημιουργία οικονομικών συνδικών όπου υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση για απασχόληση. Επομένως θα πρέπει να αδράξουμε και τις οικονομικές ευκαιρίες και προκλήσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Όλα αυτά είναι λοιπόν θετικά. Αλλά εν γέννη έχουμε ένα πιο γενικό και ίσως λιγότερο συνεκτικό ε, πλαίσιο κατευθυντηριών γραμμών. Είναι σαν ένα παιδάκι που κοιτάει τη βιτρίνα ενός καταστήματος παιχνιδιών και δεν ξέρει ακόμα πολύ καλά τι θα ήθελε να πάρει. Δεν βλέπουμε ακόμα τους συγκεκριμένους στόχους που θα πρέπει να έχουμε. Εμείς ε, από την πλευρά του Κοινοβουλίου έχουμε ακολουθήσει μια διαφορετική κατεύθυνση, μια διαφορετική αντιμετώπιση θέλουμε να καταλήξουμε στα σημεία έμφασης τα οποία είναι απαραίτητα για μας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη δημιουργία περισσότερων θέσεων απασχόλησης. Και ένα από τα σημεία αυτά στα οποία χρειάζεται έμφαση είναι προφανώς το να υπάρχουν και επιμέρους στόχοι. Ξέρω ότι σε εθνικό επίπεδο παραμένουν οι αρμοδιότητε στον τομέα αυτό, αλλά οι κατευθυντήρε γραμμέ θα πρέπει να δώσουν κάποια κατεύθυνση στα κράτη-μέλη. Και εφόσον δεν μιλάμε ακόμα για υποχρεωτικέ κατευθυντήρε γραμμέ, ίσω μπορούμε να δείξουμε λίγο πιο θάρρο και να έχουμε πιο τολμηρέ κατευθυντήρε γραμμέ και επιμέρου στόχου. Επομένω, κάναμε την πρόταση μεταξύ του μέσα στο στόχο της συμμετοχής 75% στην αγορά εργασίας ηλικιακή φέτα 20 με 24% θα πρέπει κατά 90% ή να απασχολείται ή να βρίσκεται σε εκπαίδευση και κατάρταση. Αυτό νομίζω ότι είναι αρμονικό με τον στόχο του 75% γιατί ο κύριος στόχος μας είναι να παροτρύνουμε τους νέους να περατώσουν τις σπουδέ τους το ταχύτερο δυνατό και μετά να μπουν στην αγορά εργασίας με τον τρόπο αυτό αυξάνοντας το ποσοστό απασχόλησης. Αν λοιπόν δεν μπορούμε να έχουμε ένα συγκεκριμένο στόχο εκεί, χάνεται η ορμή και η παρότριση. Κατά τα άλλα το 75% παραμένει. Επίσης, στην κατευθυντήρια γραμμή υπαριθμών 10 αναφέρθηκα στο θέμα της ένδυας των παιδιών. Ξέρουμε ότι τα παιδιά τα οποία θίγονται από την ένδυα έχουν μικρότερες ευκαιρίες στην ε, παιδεία και στην αγορά εργασίας. Και θα πρέπει να ληφθεί αυτό υπόψη για να υπάρξει και μεγαλύτερη απασχόλησή τους. Εγώ θα ήθελα να το αναφέρω και αυτό μέσα σε μια τροπολογία, να τονίσω και τη σημασία της ισότητας των φίλων και τη συμμετοχή τόσο των νέο ναι, τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών στην αγορά εργασίας. Κάτι τέτοιο όμως μπορεί να ευδοκιμήσει μονάχα αν η παιδική σταθμή που η βρεφική και παιδική σταθμή όπου είναι τα παιδιά όταν οι μητέρες τους εργάζονται θα πρέπει να έχουν τέτοιο χαρακτήρα που να επιτρέπουν στις ε, μητέρες να εργάζονται πλήρως και να έχουν συγχρόνω την εμπιστοσύνη ότι υπάρχει σωστή φροντίδα των παιδιών τους από αυτούς τους φορεί. Το Συμβούλιο επίσης δεν έχει αντιδράσει <clears throat> σε κάτι το οποίο μισθέσαμε σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, ότι αλλάζει και η φύση τη εργασία μορφή και αυτό συμβαδίζει φυσικά με, την, ε, με τις μεταλλαγές στην οικονομική δραστηριότητα, η ανάδυση μη συμβατικών μορφών απασχόλησης, για τις οποίες δεν νομίζω ότι εμείς παρέχουμε επαρκείς κατευθυντήριες γραμμές. Έχουμε τα λέτε, τις λεγόμενες ατυπικές συμβάσεις που σιγά σιγά αντικαθιστούν τις ε, συμβάσεις αορίστου χρόνου, έχουμε συμβάσεις μερικής εργασίας, έχουμε ένα ευρύτατο φάσμα εναλλακτικών μορφών εργασίας, των οποίων και η νομική ρύθμιση ελείπει ή υπάρχει σε πολύ χαμηλό επίπεδο σε πολλά κράτη-μέλη και τονίζουμε ότι για να μπορέσουμε να αυξήσουμε τη σημασία των θέσεων εργασίας ατυπικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρεται κάτι και στις κατευθυντικές γραμμές μας ώστε τα κράτη-μέλη να μην έχουν ε, αποκλίνουσες νομοθεσίες σε σχέση με την ατυπική εργασία. Σήμερα το πρωί λοιπόν συζητήσαμε μια έκθεση για ατυπική εργασία ήδη στην Επιτροπή μας και υπάρχει μια διαμάχη σε σχέση με την εκπαίδευση είτε στο σχολείο είτε εκτός σχολείου γιατί εκεί ο στόχος μας θα πρέπει να είναι η εκπαίδευση εκτός σχολείου, οι μαθητείες να έχουν ένα χαρακτήρα απόκτησης προσόντων που ευνοούν την κατάληψη θέσεων απασχόλησης. Και οι στόχοι της συνοχής θα πρέπει, μάλλον τα κονδύλια της συνοχής θα πρέπει να εξυπηρετούν τους στόχους της απασχόλησης Ιδίως μέσα στα πλαίσια της τωρινής κρίσης. Γιατί η κρίση αυτή δεν έχει μειώσει, αντίθετα έχει οξύνει τις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τα ποσοστά απασχόλησης. Επομένως, μέσα στην εργαλειοθήκη μας θα πρέπει να περιλάβουμε και τα μέτρα τα οποία θα προσπαθήσουν να εξαλείψουν αυτές τις διαφορές. Προσπαθούμε λοιπόν να δούμε πού υπάρχουν αποθέματα και μέσα σε αυτά περιλαμβάνονται και τα από θέματα για τον χώρο της εργασίας. Είναι και οι άνθρωποι με αναπηρίες. Είναι σημαντικό να δώσουμε μια μεγαλύτερη έμφαση για τα άτομα αυτά. Θα πρέπει να προσαρμόσουμε λοιπόν τις δυνατότητες απασχόλησης και στις ανάγκες αυτών των ατόμων, τότε θα μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε ένα μεγάλο αριθμό από εργοδότες, οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν στα άτομα αυτά ευκαιρίες. Εν κατακλείδη. Πιστεύουμε ότι το να υπάρχουν πιο εξειδικευμένοι επιμέρους στόχοι οι οποίοι θα θεσπιστούν θα ήταν θετικό. Γι' αυτό εγώ σας τονίζω το στόχο 90% εκπαίδευσης, κατάρτισης ή απασχόλησης για τους νέους. Το να υπάρξει επιστημονική... Οι επιστημονικές έρευνες μάλιστα λένε ότι αυτό είναι πολύ χαμηλό ποσοστό και λένε ότι οι νέοι σε αυτή την ε, ε, φέτα ηλικία θα έπρεπε να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή στην εκπαίδευση. Αυτό λοιπόν θα είναι μια προϋπόθεση για να μπορέσουν να μπουν επιτυχώς στην αγορά εργασίας και θα πρέπει επίσης να αντιδράσουμε στις μεταβαλλόμενες ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο χώρο της ε, απασχόλησης και της αγοράς και η πολιτική συνοχής θα πρέπει να παίξει και ένα ενσωματικό ρόλο για όλους αυτούς και φυσικά είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε ότι οι προτάσεις μας είναι οι βέλτιστες για να επιτεθεί μια λύση και εγώ είμαι διαθέσιμο να το συζητήσω αυτό με όλους τους ενδιαφερόμενους. Θα πρέπει να υπάρξουν φυσικά παράλληλα και οικονομικές κατευθυντήριες γραμμές ή ίσως μέσα σε κάποιο οριζόντιο <clears throat> φόρουμ μπορούμε να συνδυάσουμε τις προτάσεις απασχόλησης και οικονομικής δραστηριότητας ώστε να καταλήξουμε σε λύσεις οι οποίες δεν θα είναι μόνο θεωρητικές στον τομέα της απασχόλησης αλλά θα συνδέονται και με άλλους τομείς που έχουν επίπτωση στην απασχόληση και φυσικά ο κύριος στόχος μας θα είναι να λειτουργήσει ο στόχος του 2020, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό θα εξυπηρετηθεί από τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και να βγούμε και από την τωρινή κρίση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να δώσω τώρα το λόγο στους υπόλοιπους από τον ζήτηση κυρία Στάινρουκ. Θα σας παρακαλέσω να μην μακρηγορήσετε κι εσείς τόσο πολύ. Ευχαριστώ κύριε Κροκέτ, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και για την παρουσίαση που κάνετε των κατευθυντήριων γραμμών. Έχουν καλυφθεί ορισμένα θέματα ήδη σε επίπεδο περιεχομένου, γιατί έχουμε συζητήσει ήδη στην Επιτροπή μας για τα θέματα αυτά, τα κύρια ζητήματα, γι' αυτό εγώ δεν θα είμαι εκτενής. Νομίζω ότι ήδη γνωρίζετε ποιε είναι οι κατευθυντήριες γραμμές που θέλουμε εμείς να τονίσουμε, η παρουσία των νέων στην αγορά εργασίας, το θέμα της ποιότητας εργασίας, όλα αυτά είναι πολύ προσφυλή στην Επιτροπή μας. Εγώ όμω ζήτησα το λόγο γιατί θα ήθελα να σταθώ στο θέμα του χρονοδιαγράμματος και της συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή τη διαδικασία. Οι πολίτες της Ευρώπης μας έχουν εκλέξει για να εκπροσωπήσουμε τα συμφέροντά τους. Και εγώ ως σκιώδης εισηγητρία έχω να αντιμετωπίσω το θέμα αυτό. Εφόσον λοιπόν το θέμα αυτό θα αντιμετωπιστεί σύντομα, τον Ιούνιο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και εμείς επίσης θα ψηφίσουμε το Σεπτέμβριο, νομίζω ότι θα πρέπει να έχετε υπόψη στο γεγονός ότι η θέση της Επιτροπής Παπασχόλησης είναι πολύ κοντά στη φωνή των πολιτών. Είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη και από το Συμβούλιο η άποψη της Επιτροπής Απασχόλησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας παρακαλώ λοιπόν κατεπηγόντως να μην κλείσει τη θέση του το Συμβούλιο τον Ιούνιο, αλλά να λάβει υπόψη τη δική μας άποψη, γιατί οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι αυτοί οι οποίοι είναι πιο κοντά στους πολίτες και θα πρέπει να συζητήσουν με αυτούς και επομένως θα πρέπει η απόφαση του Συμβουλίου να λάβει υπόψη και την, τις προτάσεις που έρχονται από τους απλούς πολίτες από την Ευρώπη μέσω ημών. Τούρουναν και Κορνέλσεν μετά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Κροκέ που ήρθατε να μας μιλήσετε σήμερα. Θα ήθελα δύο πράγματα να πω. Πρώτα απ' όλα, η συνθήκη βάση για την κατευθυντήρια γραμμή υπαριθμών 10 και εσείς το σχολιάσατε και εγώ κοίταξα τη βάση τη νομική στη συνθήκη και είναι σημαντικό όλα αυτά να είναι σωστά. Εάν λοιπόν θέλετε τη δική μου γνώμη για τον κοινωνικό αποκλεισμό, η βάση που έχει αναζητηθεί στη συνθήκη είναι το άρθρο 3. Και εδώ σας παραθέτω το κείμενο της συνθήκης. Καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και τα λοιπά. Και, τα λοιπά. και στο συνθήκη του TFTU στο άρθρο 9 λέγεται ότι στην εφαρμογή των κοινωνικών της πολιτικών η Ένωση πρέπει να λάβει υπόψη τις απαιτήσει για να εξασφαλίσει υψηλά επίπεδα κοινωνικής προστασίας, απασχόλησης και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού. Στη συνθήκη ούτως ή άλλως υπάρχουν και άλλα άρθρα που προσφέρονται ως δεχόμενη νομική βάση. Θέλαμε λοιπόν σε αυτή την Επιτροπή ε, να μα πείτε κατά πόσον συζητήθηκε στο Συμβούλιο νομική βάση αυτή που μπορεί να αναζητηθεί στη συνθήκη. Εμεί πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να ισχύσει. Και αυτό μα απασχολεί. Η καταπολέμηση τη ένδυα στην Ευρώπη, οι συνθήκε διαβίωση των εκατομμυρίων που ζουν σε συνθήκε φτώχεια, των φτωχών μισθωτών. Αυτό είναι κάτι που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε και ένα μήνυμα από τη δική μα την Επιτροπή θέλουμε να αποσταλεί για το θέμα αυτό προ τον έξω κόσμο επίση οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση και την, ε, τις κοινωνικές υποθέσεις και πώς αυτές συνδυάζονται. Λέτε ότι χρειαζόμαστε συγκεκριμένα πολιτικά εργαλεία για να δημιουργήσουμε θέσει εργασία. Σωστά. Συμφωνώ. Αλλά το σημείο αφετηρία μα ποιο θα είναι. Μόνο οι περικοπέ ε, και οι περιορισμοί στου προπολογισμού, πώ θα συνδυαστούν αυτά, πώ θα συνδυαστεί η οικονομική ανάπτυξη με την απασχόληση, πώ θα μα πάρουν στα σοβαρά για του κοινωνικού μα στόχου. Η ε, ενοποίηση λοιπόν των προπολογισμών από αυτή καθεαυτή μπορεί να είναι επικίνδυνη για την αύξηση των θέσεων απασχόληση. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει βούληση πολιτική, να επενδύσουμε στι σωστέ κατευθύνσει. Θα ήθελα λοιπόν τα δικά σα σχόλια για αυτό το θέμα, να δούμε τι θα μπορούσαμε να αναλάβουμε κι εμεί ω δράση. Ευχαριστώ. κυρία Κον Έλισον, σας ευχαριστούμε για την προσελευσή σας. πολύ σωστά τονίσατε ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθούν θέσεις εργασία. Θέλουμε να προετοιμάσουμε τους ανθρώπους, να τους εκπαιδεύσουμε, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και θέσει εργασία που να μπορούν να πληρωθούν από αυτού. Και επίσης δεν ε, ικανοποιήθηκα ιδιαίτερα για να άκουσα να αναφέρετε τις πράσινες θέσει εργασία. Αν θέλουμε να πετύχουμε του στόχου τη Ευρώπη το 2020, δηλαδή να δημιουργήσουμε οικονομία πράσινη, ευθύη και συμμετοχική, τότε οι επενδύσεις στις πράσινες θέσεις εργασίας είναι απαραίτητες. Επίσης, οι οικολογικές αυτές τις εργασίας πρέπει να δημιουργηθούν, αλλά θα πρέπει να δημιουργηθεί και το εργατικό δυναμικό για να τις πληρώσει τις θέσεις αυτές. Όχι μόνο τώρα, αλλά να λάβουμε υπόψη και την γύρανση του πληθυσμού. Κάτι που θα επηρεάσει περίπου σε 10 χρόνια την ε, κατάσταση της αγοράς εργασίας πολύ σοβαρά. Επίσης, πρέπει να σκεφτούμε τις εργασιακές διευθετήσεις. Πολλής λόγος γίνεται για το συνδυασμό της περίθαλψης και της εργασίας, να υπάρχει περισσότερη ευελιξία για τους εργαζομένους. Όμως, διερωτώμεθα, πόσο μακριά τα κράτη-μέλη μπορούν να πάνε προκειμένου να επιφέρουν τις απαραίτητες αλλαγές. Λόγω χάρη, στο να προσφέρουν ε, στους ανθρώπους το δικαίωμα στην ε, εργασία μερικής απασχόλησης, ευέλικτα ωράρια και επίσης μέρος της ε, μερικής αυτή εργασίας να μπορούν να την φέρουν εις στο σπίτι τους για να μπορούν να συνδυάσουν και το χρόνο που πρέπει να αφιερώσουν στα παιδιά τους, το σχολείο των παιδιών με την εργασία. Ε, εδώ θα ήθελα την άποψή σα, γιατί οι ατυπικέ εργασίε μπορεί να καταλήξουν να γίνουν τυπικέ και αυτέ, κλασικέ και συνηθισμένε. Και το αν θα χάνουμε κόσμο από την αγορά εργασία, αυτό θα εξαρτηθεί από το αν μπορούμε να συνοδεύσουμε ε, τα δικαιώματα των εργαζομένων ε, με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται και με την κοινωνική τους προστασία, την κοινωνική περίθαλψη. Τώρα για την ευελιξία και ασφάλεια. Το θέμα είναι να δημιουργήσουμε ένα ευέλικτο σύστημα εμείς που να παρέχει και την ασφάλεια και μετά την ευελιξία. Θα προτείνουμε λοιπόν τροπολογίες για να συμπεριληφθεί και αυτή η προτεραιότητα και απλώς θα θέλαμε τα πρώτα σας σχόλια, τις απαντήσεις σας αυτά. Ευχαριστούμε. Καθότι οι ώρες έρχονται τρόχοντας, έχουμε τώρα εννέα αγορητές που ζητούν το λόγο. Θα σας αναγκάσω βεβαίως να περιορίσετε το χρόνο ομιλία σας, διότι θα ζητήσω και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τοποθετηθεί ως προς το χρονοδιάγραμμα. Αλλά όσο ήθεστε, θα γίνει αυτό μετά τις παρεμβάσεις των αγορητών μας. Και ο κύριος ε, Ροκέ ελπίζουμε ότι θα έχει το χρόνο να απαντήσει σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Η κυρία Σρέτερ και μετά η κυρία Ράπτη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Ένα κεντρικό ερώτημα. Είπατε ότι η συγκέντρωση των προσπαθειών μας θα πρέπει να είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και εδώ ρωτούμε ποιο ρόλο παίζει η πρωτοβουλία για τις πράσινες θέσεις εργασίας, πράσινες που αναπτύσσεται από το Κοινοβούλιο με τη δική μου έκθεση. Δεύτερον, αυτό που λέτε είναι ότι η κοινωνική ενσωμάτωση θα πρέπει να συνδέεται με το να δώσουμε στους ανθρώπους εργασία. Αλλά μια προϋπόθεση για αυτό το οποίο θέλετε να κάνετε είναι να υπάρξει υλοποίηση του στόχου της Κομισιόν και για την εκπαίδευση και για την περαιτέρω κατάρτιση. Δηλαδή να μπορούν να μένουν σε θέση εργασίας οι εργαζόμενοι ενώ επανεκπαιδεύονται και αποκτούν νέες δεξιότητες. Δεν πρέπει λοιπόν να ξεχάσουμε ότι για την ενσωμάτωσή τους είναι απαραίτητη η κατάρτισή τους. Γιατί δεν υποστηρίζετε περισσότερο αυτό το στόχο. Η κυρία Ράπτη και ο κύριος Πουπάκης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, θέλω να πω πρώτα ότι καλύφθηκα απολύτως από την τοποθέτηση της ε, σκιώδους εισηγήτριας των σοσιαλιστών της κυρία Στάινακ. Ωστόσο έχω μία σκέψη ή μία ερώτηση αν θέλετε που απευθύνεται και προς τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου αλλά και προς την Επιτροπή μας και προς καθέναν από εμά. Διάβασα με όση περισσότερη προσοχή μπορούσα το θέμα της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Ε, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω την έκφραση ότι έχω κουραστεί εντός εισαγωγικών να ακούω συνέχεια συζήτηση για την Ευρώπη του 2020. Γιατί? Γιατί όσο εμείς συζητάμε για την Ευρώπη του 2020, φαίνεται ότι η Ευρώπη του 2020 έχει ήδη πεθάνει εντός εισαγωγικών. Μιλάμε για νέες θέσεις εργασίας, μιλάμε για εξασφάλιση, μιλάμε για ασφάλεια, μιλάμε για προοπτικές, μιλάμε για ποιοτικές θέσεις εργασίας και την ίδια στιγμή η οικονομική πραγματικότητα που αγγίζει την Ελλάδα, που αγγίζει την Ισπανία, που αγγίζει την Πορτογαλία, που αγγίζει τη Βρετανία, μας φέρνει αντιμέτωπους ως Ευρώπη με μια νέα πραγματικότητα που λέει ότι γίνονται πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα για την είσοδο των νέων στην αγορά εργασίας, που αναγκαζόμαστε ε, να βλέπουμε μισθούς να μειώνονται συνεχώς και να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα και που αναγκαζόμαστε το κάθε κράτος χωριστά για να είναι στο πλαίσιο μιας ρεαλιστικής προσέγγισης να προσαρμόζουμε τους εθνικούς στόχους σε ένα πλαίσιο που να λαμβάνει υπόψη τις ειδικές συνθήκες κάθε κράτους μέλους. Θέλω η Ευρώπη του 2020 να πετύχει. Θέλω οι ποσοτικοί στόχοι να επιτευχθούν. Μόνο που πραγματικά, μιλώντας ειλικρινά, δεν βλέπω το δρόμο. Μιλάμε για πράσινες θέσεις εργασίας, μιλάμε για λευκές θέσεις εργασίας, αλλά δεν μιλάμε για αυτό που όλοι έχουμε στο μυαλό μας και το βλέπουμε, για το μαύρο μέλλον που πρέπει να το φωτίσουμε για την νεολαία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Να θυμίσω απλώ του συναδέλφου ότι η συζήτησή μα αφορά κυρίω τι κατευθυντήριε γραμμέ. Είναι βεβαίω ευκαιρία να αναφερθούν και άλλα θέματα μαζί. Διότι έχουμε μπροστά μα μια τάμπουλα ράζα κατά κάποιο τρόπο. Και έχουμε την πρόταση των συγητών, την πρόταση τη Επιτροπής... Ίσως καλό θα ήταν να επικεντρωθούμε και στις τροπολογίες που θέλαμε να επιφέρουμε στο κείμενο, τα κείμενα που έχουμε μπροστά μας, επιτάπητος και να μην επιδοθούμε σε γενικότερη συζήτηση, όπου ο καθένας θα μπορούσε να συνεισφέρει κατά τις απόψεις του βεβαίως. Ας είναι η συζήτησή μας λίγο πιο συγκεκριμένη, να επικεντρωθεί στους στόχους και την πρόοδο της όλης συζήτησης και της επικοινωνίας μας με το Συμβούλιο. να επεξεργαστούμε τα στοιχεία που μας προσέφερε η ΕΜΚΟ στο έγγραφο αυτό που απεστάλλει και στο Συμβούλιο και τις συγκεκριμένες προτάσεις του εισηγητή μας. Ο κύριος Πουπάκης και μετά κυρία Τσιμέρ. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Συμφωνώ με το πνεύμα της πρώτης Επιτροπής, αλλά θα ήθελα και προφορικά και μέσα από τις τροπολογίες, για αυτές θα αναφερθώ, να δοθεί μια ιδιαίτερη σημασία επιγραμματικά σε ορισμένα σημεία. Δηλαδή, στο απαραίτητο της υιοθέτηση της μελλοντική πολιτικής για την απασχόληση που πρέπει να ληφθούν υπόψη τα διαφορετικά σημεία εκκίνηση των κρατών μελών. Δεν είναι για όλους. Σημαντικό επίσης να οθεί επιπλέον βαρύτητα στην ποιοτική διάσταση της απασχόλησης, στην ουσιαστική ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου και τη διαφύλαξη του θεσμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων που αυτή τη στιγμή καταστρατηγούνται. Να γίνει σαφής αναφορά στην δημιουργία θεσμικού πλαισίου ρύθμιση των άτυπων μορφών απασχόλησης, και τη διασύνδεσή τους με ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Παράλληλα βέβαια με την ενίσχυση των ελεκτικών μηχανισμών για την καταπολέμηση της μαύρης αδήλωτης εργασίας. Στόχο μας πρέπει να είναι η πλήρης και σταθερή απασχόληση. Και τέλος, ένας ουσιαστικός συντονισμός τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση της οικονομικής στρατηγικής με τη στρατηγική απασχόλησης για να ενδυναμωθεί η κοινωνική συνοχή που είναι απαραίτητη, να λειτουργήσει αποτελεσματικά και σαν παράγοντας άμβλησης των ανισοτήτων, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κυρία Τσίμερ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κροκέ που ήσασταν εδώ παρόν και μας παρουσιάσατε τα θέματα αυτά των κατευθυντηριών γραμμών. Θα χαιρόμουν όμως ακόμα περισσότερο αν λαμβανόντουσαν υπόψη και οι προτάσεις και οι διατυπώσεις της δικής μας Επιτροπής. Είπατε ότι το Εαρνό Συμβούλιο δεν κατέληξε κάποιους στόχους για την καταπολέμηση της ένδυας. Αυτό σημαίνει ότι είναι ακόμα πιο σημαντικό οι κατευθυντήριες γραμμές να περιλάβουν και το δικό μας αίτημα από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υπάρξει μια ε, κριτική για τον μέχρι στιγμής ασαφή στόχο σε ό,τι αφορά την υλοποίησή του της καταπολέμησης της ένδειας, Να υπάρξει λοιπόν επίσης και κάποια <clears throat> περαιτέρω διευκρίνηση και προβληματισμό σε σχέση με το τι ακριβώς περιλαμβάνει η ένδεια, τι σημαίνει η ένδεια να μπορούμε να βρούμε και άλλα κριτήρια ένδυας και όχι μονάχα τα παραδοσιακά οικονομικά κριτήρια. Θα ήταν πολύ σημαντικό αυτό και επίσης κάτι άλλο το οποίο εμείς θα θέλαμε να ξέρουμε είναι σε ποιο βαθμό η υλοποίηση των εθνικών στόχων μπορεί να επηρεαστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι απλώς στο τέλος να υπάρξει ένα αριθμητικό άθροισμα των προσπαθειών των κρατών μελών που θα παρουσιαστεί ως επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε κύριε Βιλ και μετά κύριε κυρία Είναι σαφέ ότι πρώτα απ' όλα είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε θέσει εργασία με ποιότητα, με υψηλή προσθέμενη αξία. Αυτό είναι και ο λόγο για τον οποίο νομίζω ότι είναι απαραίτητο η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποστηρίξει και την τροποποίηση των δομών της οικονομίας. Εν γέννη, οι θέσεις απασχόλησης οι οποίες έχουν χαθεί κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης δεν θα επαναδημιουργηθούν στο ίδιο επίπεδο. Επομένως πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την αλλαγή και συγχρόνως. Θα πρέπει να αναφερθούμε στο γεγονός ότι η πολιτική απασχόλησης θα πρέπει να εγγυάται στους εργαζόμενους τη δυνατότητα να αλλάζουν τομέα απασχόλησης και την προσαρμογή στις μεταλλαγές της αγοράς εργασίας. Και επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τους μακροχρόνιους στόχους παράλληλα με τις αλλαγές οι οποίες λαμβάνουν χώρα στην αγορά μέσα στην εκπόνηση των προτάσεών Σε ό,τι αφορά τώρα τον αγώνα κατά της ένδυας, αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρόκληση. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τη δυνατότητα σε όλες τις ομάδες του πληθυσμού να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας ανεξάρτητα από την γεωγραφική περιοχή στην οποία ζουν και ανεξάρτητα από το επίπεδο παιδείας τους. Πρώτα απ' όλα όμως θα πρέπει να τους εξασφαλίσουμε την ασφάλεια στην απασχόληση και την παροχή των απαραίτητων κινήτρων για να θέλουν και να μπορούν κιόλα να εργαστούν. Μία ακόμα παρατήρηση, η οποία αναφέρεται περισσότερο στον εισηγητή. Σήμερα είναι πολύ δύσκολο να συγκρίνουμε την κατάσταση της απασχόλησης στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν κράτη-μέλη όπου οι άνεργοι είναι αυτοί, καταγράφοντας άνεργοι μόνο αυτοί οι οποίοι παίρνουν επιδόματα ενεργείας, αλλά υπάρχουν και άνεργοι οι οποίοι δεν παίρνουν πια επιδόματα, γιατί οι χώρες έχουν ένα χρονικό όριο, 6 μήνες ή 9 μήνες για την παροχή επιδομάτων ανεργίας. Βλέπετε ότι είναι πολύ πίκυλη λοιπόν η κατάσταση και θα μπορούσε κανείς να πει ότι εκεί που είναι πιο σύντομη, σύντομο το διάστημα ε, παροχής ε, επιδομάτων είναι καλύτερη κατάσταση, όσο στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου έτσι. Κύριε Φιγερέιδο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα, ήθελα να ξεκινήσω από το σημείο που ξεκίν... όπου σταμάτησε η κυρία Ράπτη. Γιατί έχει απόλυτο δίκιο. Εδώ συζητούμε προσανατολισμούς για την απασχόληση. Αλλά αμελούμε την πραγματικότητα όπως τη ζουν οι χώρες μας, η Πορτογαλία, η Ελλάδα, η Ισπανία, όπου επιβάλλονται πολιτικές λιτότητας περικοπές στις δημόσιες επενδύσεις, αύξηση των ε, φόρων και μείωση των μισθών. Μείωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, λιγότερη εσωτερική αγορά, λιγότερες επενδύσεις, άρα λιγότερη απασχόληση, άρα περισσότερη ανεργία. Τι τις συζητάμε λοιπόν αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές και τους προσανατολισμούς. Εφόσον δεν βλέπουμε τις μακροοικονομικές πολιτικές να παρα... να αποτρέψουν από την αύξηση της ανεργίας. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα καθοριστικής σημασίας. Αυτό θα πρέπει να είναι η βάση της συζήτησή μας, το να διατηρούμε προσανατολισμούς και να παρακολουθούμε σχολαστικά την τήρηση του Συμφώνου Σταθερότητας, ενώ τα κριτήρια σύγκλησης ε, ακολουθούνται κατά αυτόν τον τρόπο, όλα αυτά διακυβεύουν ήδη τη συζήτηση που κάνουμε εδώ στο γενικότερο πλαίσιό τη για τι κατευθύνε γραμμέ ε, για την απασχόληση. Επίση, να πω ότι υπάρχουν τουλάχιστον τρία σημεία στα οποία πρέπει, τα οποία πρέπει να δούμε με προσοχή Λόγω χάρη η ευελιξία και η ασφάλεια μπορεί να σημαίνουν περισσότερη προσωρινότητα, περισσότερε επισφαλεί θέσει για του εργαζομένου. Θα σημαίνει ότι θα πρέπει ο καθένα να αποδέχεται ό,τι να είναι προκειμένου να εργαστεί και να κερδίσει κάποια χρήματα. Σε μια δεύτερη φάση, το θέμα τη ισότητα. Οι γυναίκε πλήττονται κατεξοχήν εδώ από την ανεργία, από τη φτώχεια. Η προσωρινή εργασία των γυναικών συνεχώς ε, αυξάνεται αριθμητικά στην Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να παρουσιάσουμε στόχους για να μειώσουμε την φτώχεια. Αλλά πώς θα το καταφέρουμε εάν στους προσανατολισμούς αυτούς τους μακροοικονομικούς μας, μακροοικονομικούς μας μάλλον, δεν προβλέψουμε μια βάση για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες. Αυτό θα πρέπει να είναι το βασικό ερώτημα που να απασχολήσει τη συζήτησή μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Ρενιά και η κυρία Μπλινκεβιτσιούτε. Ευχαριστώ. Μετά από αυτά που είπε η προλαλήσεσα, ναι πάντα τις κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να τις βλέπουμε μαζί με την κρίση. Και εδώ θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση για την κατευθυντήρια γραμμή 1 Βλέπω ότι είναι πολύ σημαντικό θέμα η κοινωνική σταθεροποιητές αυτόματη. Θα θέλαμε πιο σαφείς σχέσεις εδώ και όσον αφορά την κατευθυντήρια γραμμή 7. Μιλάμε για δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Δεν υπάρχει όμως ε, κάτι συγκεκριμένο όσον αφορά τον χρόνο απασχόλησης και την ε, κατάτμιση του χρόνου απασχόλησης. Και γι' αυτό θα με ενδιαφερόταν πάρα πολύ ποια θα ήταν η δική σας πρόταση σε σχέση με το... Τις περιβολικές περορίες. Λικεβίτσιουτε και Χέλμερ. Ευχαριστώ κύριε Κροκέ για την παρουσία σας. και για τη δυνατότητα που μας δίνετε να συζητήσουμε μαζί σας. Δύσκολο να αμφιβησβητήσουμε την αναγκαιότητα αυτών των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση. Είναι καλό να υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές, όμως εμφανίζεται ένας κίνδυνος εδώ. Δεν πετύχαμε τους στόχους της Λισαβόνας. Θα πετύχουμε τους στόχους των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση. Ο στόχος είναι φιλόδοξος. Περνάμε από το 70% στο 75% απασχόληση του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Πολύ φιλόδοξος στόχος. Για την φτώχεια. Κατευθυντήρια γραμμή 10. Μειώσαμε το στόχο μας. Αρχικά μιλούσαμε για εξάλληψη της φτώχειας, ειδικά της παιδικής φτώχειας. Τώρα μετριάζουμε τους στόχους μας. Θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε τα ποσοστά απασχόλησης για να μειώσουμε τη φτώχεια και τα 20 εκατομμύρια άτομα παραδείγματο χάρη. Θα ήθελα να μάθω ποιοι θα είναι οι μηχανισμοί και τα μέσα που θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουμε ώστε τα κράτη-μέλη που ενδιαφέρονται για την εφαρμογή των κατευθυντήρων γραμμών, ειδικά όσον αφορά την καταπολέμηση της φτώχειας, να μπορέσουν να το κάνουν. Να σας πω όμως ότι ειδικά στη χώρα μου δεν υπάρχει πολιτική βούληση για καταπολέμηση της στόχιας. Και εδώ δεν μιλάμε απλά για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Πρέπει να βρούμε με τη βοήθεια και του Συμβουλίου και της Επιτροπής τα μέσα που θα μας επιτρέψουν να επιτύχουμε την εξάλληψη της φτώχειας. Μετά, μηχανισμοί καταπολέμησης της μαύρης εργασίας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι που εργάζονται μαύρα. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Ευχαριστούμε κύριος Λεμέρ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Άκουσα τη συζήτηση αυτή με ιδιαίτερη προσοχή και Πράγματι και σε σχέση με τα προηγούμενα σημεία της συζήτησής μας το πρωί βρίσκω ότι η συζήτηση αυτή έχει να, κάνει, έχει να μας απασχολήσει πολύ. Εδώ το θέμα είναι να δούμε τι θα γίνει βεβαίως και με τα θέματα αυτά και πώ θα έχουμε τι σωστέ προσδοκίε και στόχου. Βεβαίω θέλουμε να μειώσουμε τη φτώχεια και την ε, ανεργία των ε, νέων. Αυτή όλοι οι στόχη είναι πολύ θεμητοί. Αλλά αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε είναι με δύο κουβέντε στο νόημα των κατευθυντήριων γραμμών. τα πάμε όλοι καλύτερα. Αλλά το θέμα είναι πώ ακριβώ θα γίνει αυτό και πώ θα το πετύχουμε. Βεβαίω ότι οι συνάδελφοι εδώ ε, κινητοποιούνται από πραγματική συμπόνια για του ε, συμπολίτε οι οποίοι έχουν σοβαρέ δυσκολίε. Όμω, στο βαθμό που δεν προτείνουμε συγκεκριμένου μηχανισμού τελικά, αυτό που κάνουμε είναι ότι επιβάλλουμε νέες υποχρεώσεις στους εργοδότες να αυξήσουν το κόστος της κάθε θέση εργασίας, να μειώσουν την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών οικονομιών και οι συνέπειες αυτού, εάν ακολουθηθεί αυτή η πολιτική, είναι μικρότερη οικονομική αύξηση και μεγαλύτερη ανεργία. Άρα η συμπόνια για τους ανέργους δεν μας οδηγεί σε περισσότερη απασχόληση και περισσότερη ευημερία για τις ε, κοινότητές μας συνολικά. Εδώ θα πρότεινα, παρόλο που έχω μια αρνητική εικόνα των πραγμάτων, ότι υπάρχουν ε, και κάποιες καλές ειδήσει. Δηλαδή, να απασχοληθούμε και με το κατά πόσον εδώ κάποιος μας ακούει, αν ασχολούνται οι άνθρωποι με αυτά που λέμε εδώ μέσα λένε κάποιοι ότι οι εκθέσει γράφονται για να πεταχθούν στον κάλαθο των αχρήστων. Το είπε μια συνάδελφο. Καταλαβαίνω γιατί το σκέφτεται. Κάποιο άλλο σχολίασε ότι η επιτροπή αυτή είναι πολύ κοντά στου πολίτε. Να ρωτήσω εγώ πότε βγήκαμε και μιλήσαμε στου ανθρώπου, μιλήσαμε στου επιχειρηματίε, μιλήσαμε στου εργοδότε. Για ρωτήστε του, γιατί εκείνοι δεν μα είπανε μπράβο που δημιουργήσαμε, δημιουργήσαμε ένα περιβάλλον για να αυξηθούν οι θέσει εργασία. Μα ρωτάνε γιατί μα ε, ζαλίζεται με νέους κανονισμούς και περισσότερους κανόνες που και πολύ δύσκολοι είναι και πολλά κοστίζουν για να υλοποιηθούν και εμποδίζουν τις περισσότερες επενδύσεις και την ε, πρόσληψη νέων ε, εργαζομένων. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνουμε πρόεδρε είναι να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μικρή, λίγα πράγματα που μπορεί να κάνει το Κοινοβούλιο τελικά για να δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας αλλά πολλά μπορεί να κάνει για να άρει την έλλειψη κινήτρων για να δημιουργηθούν θέσει εργασία. Δυστυχώ στην Επιτροπή αυτή φαίνεται να είμαστε αποφασισμένοι να δημιουργήσουμε νέα αντικίνητρα για την δημιουργία θέσεων εργασία. Το αντίθετο από αυτό που θα πρέπει να κάνουμε στι δυσχερεί αυτέ τι συνθήκε τι οποίε ζούμε. Χρειαζόμαστε λιγότερου κανόνε, λιγότερη φυρολογική πίεση για να έχουμε μεγαλύτερη οικονομική αύξηση, περισσότερη απασχόληση, περισσότερε θέσει εργασία και τα υψηλά επίπεδα που όλοι αποζητούμε. Ευχαριστούμε συνάδελφε για αυτήν την ε, εκαθαριστική πρόταση. Να δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Κώστα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για αυτήν την συνάντηση. Ελπίζω ότι για όλους είναι επικοδομητική, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότως ή άλλως ότι τους προσανατολισμούς αυτούς πρέπει να τους επεξεργαστούμε και να τους συνδυάσουμε βεβαίω με την οξύτερη οικονομική κρίση που γνώρισε τι τελευταίε δεκαετίες η Ευρώπη. Όλοι λοιπόν γνωρίζουμε κατά πόσον είναι εύστοχες όλες αυτές οι πολιτικές για την Ευρώπη. Και θα πρέπει βεβαίω να αισθανθούμε και το βάρο τη ευθύνη μα για να συμβάλλουμε θετικά στου στόχου αυτού. Θεωρώ ότι, όπω σωστά επεσήμανε ο εισηγητή μα, χρειάζονται κάποιε προσαρμογέ στο κείμενο τη πρόταση των προσανατολισμών, να αναφορθούν έντονα κάποιε απαιτήσει αντιμετώπιση τη κρίση, να γίνουν πιο συνεκτικέ, πιο συνδυασμένε οι πολιτικές ε, εργασίες απασχόλησης. Είναι τρία ζητήματα τα οποία συνδυάζονται και διασταυρώνονται εδώ και τα οποία δεν υπογραμμίζονται αρκετά στους προσανατολισμούς. Θα πρέπει να ενδυναμωθεί δηλαδή το πνεύμα των ε, προσανατολισμών για τις επενδύσεις στην κοινοτομία, την έρευνα και τις ποιοτικές θέσεις εργασίας. Νομίζουμε ότι η τελευταία έκθεση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη δείχνει κάτι τέτοιο. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε ότι αυτό είναι πιο σημαντικό από ό,τι στο παρελθόν. Πρέπει να υπάρχουν σοβαρέ επενδύσει στι δεξιότητε, τα επαγγελματικά προσόντα, την κοινοτομία και την έρευνα, είτε κρατική είτε ιδιωτική. Ε, το τελευταίο σημείο το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι το εξή. Συνεχίζουμε να λέμε ότι έχει αποτύχει η πολιτική τη Λισαβόνα. Δεν ξέρω αν ήταν ε, σωστή η στατικική στην αρχική τη σύλληψη και αν έφταγε αυτό το θέμα. Να οικοδομήσουμε μια Ευρώπη που να βασίζεται στη γνώση, τι δεξιότητε και την ποιότητα. Σίγουρα αυτό δεν ήταν το σφάλμα. Το σφάλμα όμω ήταν ο τρόπο που υλοποιήθηκε ίσω. Η ανεπάρκεια των στόχων που είχαν τεθεί, των ενδιάμεσων ενδεχομένων στόχων που λείψαμε. Ίσως δεν μπορέσαμε να επεξεργαστούμε παραμέτρους συγκρίσιμους και παραμέτρους συγκρίσιμες και χρήσιμες που να είναι πιο αξιοποιήσιμες από ό,τι τελική αριθμητική στόχη. Να γίνει μια κριτική αποτίμηση των προτάσεων που γίνονταν καθώς και πρόβλεψη συγκεκριμένων μηχανισμών και κινήτρων και για τα διευθυντικά ταμεία. Τα διευθυντικά ταμεία πιστεύω ότι εδώ θα πρέπει να γίνει μια συνιστόσα στρατηγική σημασία για του ε, στόχου μα αυτού, για την απασχόληση και για ένα welfare, για μια ευημερία που να συνδυάζεται με μια μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά εργασία. Αυτό αφορά ολόκληρε γενιέ νέων που θα εργαστούν σε συνθήκε πολύ επισφαλεί, πολύ προσωρινέ. Θα πρέπει λοιπόν οι ετήσιε εκθέσει των κρατών μελών, αυτέ που πρέπει να εντάσσονται για την απόκρισή τους στους στόχους αυτούς των προσανατολισμών θα πρέπει να γίνει με μεγαλύτερη βαρύτητα, να είναι πιο υποχρεωτική η δέσμευση αυτή και το μέρος που εφορά την υπηκοδότησή μας με μηχανισμούς, με όργανα. Μιλάμε για την αποτυχία της στρατηγικής της Λισαβόνας πολύ συχνά. Εδώ η Επιτροπή μας θα έπρεπε να δώσει μια συνεισφορά θετική. Ιδάλλως θα παραμένουμε σε μια διάθεση ευκτική ε, σε σχέση με τους στόχους που θέτουμε μέσα από τους προσανατολισμούς των κειμένων μας. Ευχαριστούμε. Κυρία Κώστα ήταν η τελευταία παρεμβαίνουσα. Και... Επειδή το Συμβούλιο και η Επιτροπή έχουν αναφερθεί και σίγουρα έχουν να ασχοληθούν και με το θέμα του χρονοδιαγράμματος και πριν δώσουμε το λόγο και στον κύριο Κοκέ για να μας απαντήσει στις διάφορες ανησυχίες που διαφάνησαν μέσα από τη συζήτηση στην Επιτροπή μας κάποια από τα σχόλια, μέλλον από το χρονοδιάγραμμα έχει προκαλέσει και πολλές απογοητεύσεις και κάποιο άγχος. Η Ισπανική Προεδρία Επίση, εκπροσωπείται από τον κύριο Ιγνάσιο Μπερνάντο, τον πρόεδρο τη αρμόδια ομάδα εργασία στο Συμβούλιο. Θα του δώσουμε λοιπόν τον λόγο για να τοποθετηθεί, να μα εξηγήσει τη στάση που θα τηρήσει το Συμβούλιο για την υιοθέτηση αυτού του χρονοδιαγράμματο. Κύριε Μπερνάντο. Και για το θέμα του χρονοδιαγράμματο. Και αν υπάρχουν βεβαίω και άλλα σχόλια τα οποία θέλετε να κάνετε σε σχέση με τα όσα προηγουμένω αναφέρθηκαν στη συζήτησή μα, παρακαλώ. Κάντε το. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο για να διευκρινίσω ορισμένα θέματα χρονοδιαγράμματο, που βλέπω ότι δημιουργήσαν ανησυχίε στα μέλη τη Επιτροπής σα. Πρέπει να πω ότι και η Ισπανική Προεδρία υπέστη μεγάλη πίεση χρονοδιαγράμματος στο Ερνό Συμβούλιο έλαβε την απόφαση ότι από τη στιγμή που θα είχαν θεσπιστεί οι βάσει τη στρατηγικής 2020, ήδη από το Συμβούλιο του Ιουνίου να ξεκινήσει αυτή η στρατηγική. Και όπως ξέρετε, οι ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές είναι ένα απαράγραπτο στοιχείο για αυτή τη στρατηγική, μεταξύ των οποίων ένα σημαντικό ρόλο παίζουν οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. Η πρόταση της Κομισιόν βέβαια καθυστέρησε περισσότερο από ό,τι περιμέναμε, και δημοσιεύτηκε μονάχα στις 27 Απριλίου. Δηλαδή όταν είχε προχωρήσει αρκετά το εξάμεινο της Ισπανικής Προεδρίας. Παρ' όλα αυτά θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να συνεχίσουμε με την ιδέα να ξεκινήσει η στρατηγική αυτή τον Ιούνιο. Υπάρχει αυτό το χρονοδιάγραμμα. Εκπνέει η, τωρινή στρατηγική. Τα εθνικά προγράμματα θα παρουσιαστούν το φθινόπωρο και αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να αναφέρονται στις κατευθυντήριες γραμμές απασχόλησης. Γι' αυτό το Συμβούλιο, στο επόμενο Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης 7 Ιουνίου στο Λουξεμβούργο, θα προσπαθήσει να δώσει γενικές κατευθύνσεις και να επιζητήσει και την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Πάντως, η απόφαση δεν θα μπορέσει να ληφθεί παρά μόνο όταν είναι γνωστή και έχει τύχει επεξεργασία η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό θα γίνει φυσικά υπό την Βελγική Προεδρία, γιατί η ψηφοφορία για την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα λάβει χώρα το Σεπτέμβριο. Θα γίνει λοιπόν το φθινόπωρο η περαιτέρω επεξεργασία και η Βελγική Προεδρία προβλέπει στο χρονοδιάγραμμα της να εγκριθεί από το Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης τον Οκτώβριο και να περάσει μετά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου. Δεν σημαίνει ότι έχει σταυρώσει τα χέρια του και δεν κάνει τίποτα το Συμβούλιο όλο αυτό το διάστημα. Εμείς έχουμε παρουσιάσει και τη θέση μας σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν και έχουμε τροποποιήσει το κείμενο αυτό βάσει και των στοιχείων που μας έδωσε η Επιτροπή Απασχόληση και θέλω ευχαριστήσω τον Μπρούνο Κοκέ για την εργασία που έχει κάνει σε ένα πάρα πολύ μικρό διάστημα η δική του Επιτροπή για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις προτάσεις τροποποίησης που παρουσιάστηκαν από τα κράτη-μέλη και επίσης λαμβάνοντας υπόψη και προτάσεις από, άλλες, από φορεί, φορείς, χάρη την Επιτροπή Παιδεία, η οποία έκανε σχόλια για τι κατευθυντήρες γραμμέ και επίση την Επιτροπή Κοινωνική Προστασία, η οποία και αυτή έκανε προτάσει σε σχέση με την, οδηγία, την κατευθυντήρια γραμμή υπαριθμών 10. Επίσης η ομάδα εργασία για τα κοινωνικά θέματα έκανε συνεισφορές και η Οικονομική Επιτροπή και τελικά όλα αυτά μας έχουν οδηγήσει σε ένα κείμενο το οποίο διαφέρει από την, πρόταση, από την αρχική πρόταση της Κομισιόν, το οποίο θα παρουσιαστεί στο Συμβούλιο Απασχόλησης και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και πιστεύω ότι με τον τρόπο αυτό θα έχουμε συλλέξει πολλές από τις απόψεις που ακούσαμε και ε, στην συνεδρία της Επιτροπής σας στο Στρασβούργο, όπως και εδώ σήμερα. Ευχαριστούμε για αυτές τις διακριβώσεις και το τι μορφή θα πάρει η διαδικασία υιοθέτηση των εθνικών γραμμών. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν και οι συγκεκριμένε διαπραγματεύσεις μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Ίσως να παραταθούν, ίσως να οριστικοποιηθεί τελικά η θέση επί του θέματος αυτού. Κύριε Πρόεδρε, δεν θα σας έλεγα να απαντήσετε σε κάθε ένα από τα σημεία της κάθε μιας από τις παρεμβάσεις που έγιναν. Ίσως και βάσει των προτάσεων του Ισηγητού μας, να δώσετε έμφαση στα σημεία που φαίνονται πιο σημαντικό, σημαντικά για τη συνέχεια της συζήτησης μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Λαμβάνοντα υπόψη βεβαίω και τι τοποθετήσει των ΜΕΝ και των ΔΕ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ για όλα αυτά τα σχόλια και όλες τις ερωτήσεις σας. Προφανώς στην ΕΜΚΟ εργαζόμαστε βάσει των όσων μας ζητά το Συμβούλιο. Σε γενικές λοιπόν γραμμές και για να απαντήσω στις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις των εισηγητών, του εισηγητή μάλλον συγκεκριμένα, έχω δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο πνεύμα το οποίο έγιναν οι τροπολογίες μας και δεδομένου και του χρονικού πλαισίου. Δηλαδή, Συμπυκνώνοντα το πνεύμα αυτό, θα επιμείνω στο έχουν συνταχθεί κατά τρόπο ώστε να αναφέρονται όλα τα σημεία που έλειπαν και που μας φαίνονταν σημαντικά, ιδίω τα δημοσιονομικά εργαλεία, αλλά και άλλα επικοδοτήσει και το καθεξής, δεν θα σταθώ σε αυτά. Παρόλα αυτά, οι κατευθυντήρες γραμμέ τουλάχιστον επιτρέπουν να γίνουν όσα γίνονταν στο παρελθόν και κάτι παραπάνω, με τρόπο πιο σαφή για ορισμένα τουλάχιστον σημεία. Κατά τρίτον, για την σύνταξη. Δεν εμποδίζει τίποτε να κάνουμε αυτά που επιθυμούμε, ώστε να επιτύχουμε τους στόχους τους οποίους αναλάβαμε να επιδιώξουμε. Τώρα, σε σχέση με όλε αυτέ τι παρατηρήσει για την ισότητα των φύλων, για την και ασφάλεια, για του νέου και ούτω καθεξής, δεν νομίζω ότι επί της ουσίας διαφωνούμε. Και, δηλαδή εμείς και τα μέλη της Επιτροπής σας. Σίγουρα μεταξύ των κρατομελών υπάρχουν κάποιες αποκλήσεις απόψεων. Όμως συνολικά για το ποια κατεύθυνση θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Δεν φαίνεται να υπάρχει πραγματική διαφωνία το γράμμα των κατευθυντήριων γραμμών ως έχει, σαφώς ε, από κάποιες σκοπιές μπορεί να παρουσιάζει μία υποβάθμιση σχετική, από κάποια άλλη άποψη παρουσιάζει βελτιώσεις, αλλά είναι ο μόνος τρόπος να υλοποιηθούν οι πολιτικές απασχόλησής μας. Αυτό είναι και ο λόγος που είναι ικανοποιημένη η ΕΜΚΟ στο σύνολό της σε σχέση με τις τροπολογίες που επιφέρθησαν. Τώρα, για να μπορέσουμε να συνδυάσουμε την πρόταση του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, θα πρέπει να συζητήσουμε. Αυτό θα πρέπει να είναι ο στόχο μα. Δηλαδή, τι μα ενδιαφέρει να πετύχουμε με αυτέ τι κατευθυντήριε γραμμέ. Τι μπορούμε να κάνουμε και τι δεν, μπορούσαμε να, δεν μπορούμε να κάνουμε πλέον που μπορούσαμε στο παρελθόν. Ή τι μπορεί να αλλάξει. Σε σχέση με αυτέ τι προτάσει, λοιπόν, είναι πολλά τα σημεία στα, να, στα οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε. Έπειτα, σίγουρα υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Όπω εάν θα πρέπει να υπάρχουν αντικειμενικές δεσμευτικές υποχρεώσεις εδώ. Ε, σίγουρα το Συμβούλιο επέμεινε σε αυτό και το έργο της ΕΜΚΟ ήταν να επιδιώξει να έχουμε αντικειμενικές ε, αντικειμενικούς στόχους και τα, εθνικ... τα, κράτη... τα κράτη-μέλη να τους ακολουθήσουν πιστά. Θα έπρεπε λοιπόν να δούμε ποιες θα, ποιοι θα είναι αυτοί οι συγκεκριμένοι στόχοι ανάλογα με πληθυσμιακές ομάδες για να μην ξεπεράσουμε και τα όρια που προβλέπονται για τις διάφορες ομάδες και να μπορούμε να κάνουμε και σύγκριση των δεδομένων των κατομελών βάσει στατιστικής μελέτης. Αυτό ήταν ένας βασικός στόχος. Έπειτα, για το όλο πνεύμα των προτάσεων. Δεδομένου του χρόνου που είχαμε, δεν ήταν δυνατό να βελτιώσουμε την ισορροπία των κατευθυντηρίων γραμμών. Κάποιοι είπαν ότι περισσότερα μπορούσαν να γίνουν προ αυτή την κατεύθυνση, περισσότερη σαφήνεια, περισσότερε θέσει εργασία, λέγω με περισσότερη απασχόληση. Δεν είχαμε το χρόνο. Πρέπει λοιπόν να γίνει διάκριση μεταξύ του τι προέχει να φανεί μέσα από τι κατευθυντηρίε γραμμέ και τι προέχει να υλοποιηθεί μέσω τη διακυβέρνησή μα πράγματα πολύ λιγότερο επίσημα, αλλά πολύ πιο χειροπιαστά για την υλοποίηση των πολιτικών σε διάφορε χώρε. Οι διάφορε ελλείψει λοιπόν που μπορούν να υπήρχαν στο παρελθόν, μπορούν να αντιμετωπιστούν με τα νέα όργανα που προτείνονται λόγω χάρη. Για τι διάφορε προτάσει φυλάξη που αναφέρθηκαν, τι καινοτόμε πολιτικέ απασχόληση, νέα στοιχεία σε σχέση με το παρελθόν. Αλλά για όλου αυτού του στόχου το θέμα είναι πώ υλοποιούνται. Ίσως λοιπόν αυτό που προέχει εδώ δεν είναι να επιμείνουμε με κάθε τίμημα ε, στη σύνταξη του κειμένου των καθετηρίων γραμμών, αλλά να βεβαιωθούμε ότι η κυβέρνηση, η υλοποίησή τους δηλαδή, επιτρέπει να τα φέρουμε εις πέρα στα όσα προβλέπουν αυτές οι γραμμές. Αυτό είναι λοιπόν και το πνεύμα εντός του οποίου εργαστήκαμε. Έπειτα, σε ό,τι αφορά το συσχετισμό με τις μακροοικονομικές πολιτικές. Εδώ υπήρξε μια σειρά παρατηρήσεων. Πολλοί έθεσαν ερωτήματα εδώ. Βεβαίω, ο συσχετισμό με τι μακροοικονομικέ πολιτικέ είναι άκρο σημαντικό για του κοινωνικού εταίρου, για τι συμπεριλήψει που έκανε η Επιτροπή Απασχόληση στι κατευθυντήρε γραμμέ. Ε, έκανα και εγώ σχόλια. Έχουμε προτεραιότητα την εργασία. Σε αυτόν τον σκοπό συγκλίνουν όλε μα οι συμπεριλήψει. Δηλαδή, η προσφορά εργασία να μην εξασφαλίζει μόνο να προσαρμόζονται οι εργαζόμενοι στην αγορά εργασία, να υπάρχει περισσότερη διευθέτηση και κανόνε. Αυτά είναι σίγουρα σημαντικά, συνεχίζουν να υπάρχουν. Αλλά αυτό που κοιτάξαμε να διασφαλίσουμε από την άλλη είναι ότι οι μακροοικονομικές μεταρρυθμίσει επιτρέπουν τη δημιουργία θέσεων εργασία, Κάτι που δεν ίσχυε τα δέκα προηγούμενα χρόνια, λόγου χάρη, απαραίτητο. Και μεταξύ αυτών των νέων εργασιών που θα δημιουργηθούν θα υπάρχουν και πράσινε θέσει εργασία. Υπάρχει μια μνήμα εδώ, συμπεριλήφθη μια νέα μνήμα μάλιστα σε σχέση με τι προτάσει τη Επιτροπή, στι δικέ μα κατευθυντηρίε γραμμέ, όπω τι ανασυντάξαμε, και σε σημαντική μάλιστα θέση. Οι οικολογικέ λοιπόν οι πράσινε θέσει εργασία είναι ένα υποσύνολο των υπόλοιπων θέσεων εργασία και εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από τι βιομηχανικέ, μακροοικονομικέ και ούτω καθεξή πολιτικέ που σκοπό έχουν να αναπτύξουν αυτού του τομεί. Δεν θα εκπαιδεύσουμε νέους ε, για πράσινες θέσεις εργασίας αν δεν υπάρχουν θέσεις αυτές και αν δεν υπάρχει και ζήτηση για πράσινα προϊόντα. Όλε οι μελέτε που έχουν γίνει για το θέμα αυτό εγκλίνουν σε αυτό το σημείο. Αναφέρονται λοιπόν οι πράσινε θέσει εργασία και νομίζω ότι αυτό απαντά εν μέρη στι ανησυχίε σα. Και αυτέ αναφέρονται ω υποσύνολο των πολιτικών που δημιουργούν γενικότερα, γεννούν εργασία. Έπειτα, για τα σύνολα εκτό της αγοράς εργασία, τα άτομα με ειδικέ ανάγκες λόγου χάρη που αναφέρονται, τα άτομα που είναι αποκλεισμένα από το κοινωνικό σύνολο, από την αγορά εργασία. Επίση, Εδώ υπάρχουν περισσότερα από ό,τι στο παρελθόν. Οι πολιτικές όπως τώρα προτείνονται επιτρέπουν να κάνουμε περισσότερα σε ό,τι αφορά το στόχο καταπολέμηση τη φτώχεια, Η Επιτροπή απασχόληση δεν ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το στόχο αυτό, γιατί δεν είναι εντό των αρμοδιοτήτων μα των κλασικών. Η Επιτροπή τη Κοινωνική Προστασία ασχολήθηκε με αυτό το θέμα. Άλλωστε και αυτή η Επιτροπή συμβάλλει στι συζητήσει του Συμβουλίου Εύσκο οπότε είναι κοινή η ευθύνη μα και ήταν η ευθύνη του Συμβουλίου αυτού να αποφασίσει βεβαίω. Ωστόσο, στην ΕΜΚΟ, κανεί δεν θα μπορούσε να σα πει, όσου κάθισαν στο τραπέζι των συζητήσεων, ότι δεν είναι σημαντικέ και αυτέ οι πολιτικέ. Και ότι χωρί τι πολιτικέ τη κοινωνική συμμετοχή στην αγορά εργασία δεν θα καταλήξουμε στου στόχου που θέλουμε. Κανεί δεν το πιστεύει αυτό. Οι κατευθυντήριε γραμμέ όπω έχουν συνταχθεί σήμερα δεν εμποδίζουν κάτι τέτοιο. Άρα, για άλλη μια φορά, νομίζω ότι όπω και οι πολιτικέ για την ισότητα των φύλων δεν βρίσκουν ενάντια κανέναν γύρω από το τραπέζι των συζητήσεων στην ΕΜΚΟ. Κανεί δεν θα σα πει να υποβαθμίσετε τη θέση των γυναικών. Ίσα ίσα. Η σύνταξη του κειμένου μας το επιβεβαιώνουν αυτό στο γράμμα του κειμένου. Και στο πνεύμα της σύνταξής του κανείς δεν είχε τέτοια πρόθεση να ε, παραμερίσει ένα από αυτά τα θέματα ως προτεραιότητα. Έχω την εντύπωση ότι λίγο πολύ κάλυψα τα βασικά σημεία της συζήτησης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στις εργασίες μας. Ελπίζουμε ότι στη συνέχεια των εργασιών μας, εργασιών σας συγγνώμη, θα έχετε λάβει υπόψη και τις μέρημνες και τις ανησυχίες των ε, βουλευτών για το τελικό αποτέλεσμα των εργασιών της Επιτροπής σας. Ελπίζουμε ότι μπορεί να αναπτυχθεί ένα πνεύμα αγαστής συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής μας και της δικής σας. Σας ευχαριστούμε λοιπόν ιδιαίτερα για την παρουσία σας μεταξύ ημών σήμερα το απόγευμα. Υπενθυμίζω ότι για την έκθεση του κυρίου Όρη η προθεσμία κατάθεση των τροπολογιών έχει καθοριστεί για τις 4 Ιουνίου στο μεσημέρι, θα εξεταστούν στη συνέχεια στις 24 Ιουνίου. Από την Επιτροπή μας κλείσαμε το σημείο αυτό της τη διάταξης. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κρόκε. Euh, Ερχόμαστε τώρα στο σημείο 6. 6 τι λέγω στο σημείο 13 της ημερήσιας διάταξης που αποτελεί την πρώτη εξέτασή μας της ε, εκθέσεως της κυρίας Μωράν Σαρτιέ της γνωμοδότησης καλύτερα μέσα στα πλαίσια της ενισχυμένης συνεργασίας με την Επιτροπή Προϋπολογισμών σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση. Ο κύριος Πόρτας είναι ο αρμόδιος από την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Χαιρετίζω την παρουσία του και δίνω το λόγο στην κυρία Μπεθ Μωρέου Σαρτιέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης που παρουσιάζεται σήμερα για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση τοποθετείται στο ίδιο πλάνο που αφορά και το πρόγραμμα για τις ε, κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση που συζητήσαμε προηγουμένως. Να πω εδώ ότι χάρηκα πολύ για τη συνεργασία μου με τον ε, Πόρτας ε, για το θέμα αυτό, ο οποίος είναι υπεύθυνος επί της ουσίας ε, στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Πρέπει να υπενθυμίσω εδώ ότι αυτό το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση εγκρίθηκε το 2006 μετά από αίτημα του κυρίου Μπαρόζο και αφορούσε αρχικά την ανάπτυξη επενδύσεων ετέθησε επιχειρησιακή λειτουργία το 2007, αλλά είχε ελάχιστη συμμετοχή σε αυτόν το στόχο. Μετά το 2009 υπήρξε ανανέωσή του και αφορά πλέον και νέα θέματα, ενώ βεβαίως αυτή η εξέλιξη θα πρέπει να συνεχιστεί και σήμερα, καθώς βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά αιτήματα και πιο ευρύς φάκελοι πλέον. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτή την αύξηση ζήτησης με επιτάχυνση των δικών μας απαντήσεων που αυτή τη στιγμή παίρνουν 12 με 17 μήνες για κάθε αίτημα. Αυτή τη στιγμή όμως αντιμετωπίζουμε μαζικές απολύσεις και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ζουν υπό πολύ δύσκολες συνθήκες. Ένα δεύτερο θέμα. Η διερεύνηση των φακέλων σήμερα παίρνει πολύ χρόνο και θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο δραστήριοι ως Ευρώπη. Άρα όχι μόνο πρέπει να επιταχύνουμε τους ρυθμούς ε, της εργασίας μας, αλλά και να δείξουμε μεγαλύτερη δραστηριοποίηση. Τρίτον, σήμερα η χρηματοδότηση δεν ε, στοχεύει αποκλειστικά, δεν ε, προέρχεται μάλλον αποκλειστικά από το προϋπολογισμό των τακτικό, αλλά προέρχεται και από τα αποθεματικά. Όμως πρέπει να βρούμε πλέον νέες λύσεις μέσα στον προϋπολογισμό για τη χρηματοδότηση του Ταμείου. Κάτι ακόμη το οποίο θα ήθελα να τονίσω. Δεν πρέπει να παρανοούμε την έννοια του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Δεν αφορά τις επιχειρήσεις, αφορά τους υπαλλήλους την επανεισογωγή τους στην εργασία. Δεν αφορά δηλαδή προγράμματα απολύσεων των επιχειρήσεων. Και γι' αυτό θα πρέπει να εντοπίσουμε στρατηγικές επιτόπου και να εντοπίσουμε τις βέλτιστες πρακτικές που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για όλα αυτά χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες με στόχο την επανακατάρτιση του προσωπικού, την επανεισαγωγή τους στην αγορά εργασίας και δραστηριοποίηση και από τα κράτη-μέλη κάθε φορά που υπάρχουν ανακοινώσεις απολύσεων, ήδη από την ανακοίνωση. Σήμερα λοιπόν κυρία Πρόεδρε θα ήθελα να προτείνω καταρχάς να επιμείνουμε στην ανάγκη ανάπτυξης της ε, επαγγελματικής ολοκλήρωσης ως μέσου κοινωνικής ολοκλήρωσης. Τα κράτη-μέλη δεν γίνονται νονοί προστάτες. Όμως έχουμε ευθύνη απέναντι σε όλους τους εργαζόμενους για να επιτύχουμε την κοινωνική τους ένταξη. Δεύτερον, προτείνουμε να υπάρξει χρηματοδότηση σε συγκεκριμένες γραμμές του προϋπολογισμού Να εντοπίσουμε δηλαδή συγκεκριμένα μέσα προς όφελος των υπαλλήλων στα πλαίσια του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Τρίτη πρόταση, επιθυμούμε και αυτό ζήτησε και όλη η Επιτροπή ΦΕΜ, γυναικών δηλαδή, είναι να υπάρξει πραγματική δέσμευση όλων των κοινωνικών εταίρων με συγκεκριμένη διαδικασία, όχι απλά επί χάρτου, που θα διασφαλίζει ότι θα υπάρχει συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων καθ' όλη τη διαδικασία. Δεν αρκούν τα όσα ισχύουν μέχρι σήμερα. Θέλουμε μία νέα πολιτική πιο συγκεκριμένη και διαρθρωμένη. Το τέταρτο σημείο που προτείνουμε είναι ανάπτυξη της επικοινωνίας για το Ταμείο στα κράτη-μέλη και στην Ευρώπη, προκειμένου όλοι να γνωρίζουν τη διαδικασία και να μην γίνεται αυτό που συμβαίνει σήμερα, όπου Υπάρχουν κάπου 10 κράτη-μέλη που δεν έχουν προσφύγει ποτέ στο Ταμείο. Και σίγουρα υπάρχουν ανάγκες και σε αυτά τα κράτη-μέλη που δεν καλύπτονται, προφανώς επειδή υπάρχει άγνοια του Ταμείου και γιατί δεν έχει υπάρξει κατάλληλη ενημέρωση. Πέμπτη πρόταση θέλουμε να υπάρξει πολύ πιο θετική διατύπωση της δυνατότητας κάποια κράτη-μέλη να μπορούν να κάνουν κοινά αιτήματα. Είτε πρόκειται για παραμεθόριες περιοχές, είτε σε περιπτώσεις μεγάλων επιχειρήσεων. Υπήρξε μια τέτοια περίπτωση Και αν είχαμε αυτή τη δυνατότητα, θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ πιο, καλύτερα, πιο καλά αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή όμως είναι αλήθεια ότι δεν αποκλείεται η δυνατότητα καινού αιτήματο από περισσότερα κράτη-μέλη, αλλά θα θέλαμε να αναφέρεται και ρητός αυτή η δυνατότητα. Ένα ακόμη σημείο. Θέλουμε μια πιο εξατομικευμένη προσέγγιση για τους απολυμένους εργαζόμενους μέσω του Ταμείου έτσι ώστε να είναι πραγματικά αποτελεσματική η πολιτική επανένταξής τους στην εργασία. Εξατομίκευση λοιπόν για να μπορούμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Έβδομο. Αυτό το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση επιτρέπει την ε, απόκτηση νέων προσέοντων από τους απολυμένους προκειμένου να βρουν νέες θέσεις εργασίας και αυτό ναι μεν ισχύει γενικά για τη δημιουργία απασχόλησης αλλά είναι πραγματικά επίγουσο σημασίας όταν μιλάμε για απολυμένους εργαζόμενους. Πρέπει λοιπόν κάθε απολυμμένος εργαζόμενος να μπορεί να αποκτήσει μία νέα επαγγελματική καριέρα και νέες επαγγελματικές προοπτικές. Όδον, έχει να κάνει με την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων και είναι πολύ σημαντικό για εμένα γιατί θα πρέπει η όλη διαδικασία της πιστοποίησης εμπειρίας να γίνεται πριν την απόλυση, έτσι ώστε να μπορεί μετά ο απολυμένος και να μπορεί να μεταβεί εύκολα σε κάτι άλλο, αλλά και να μπορεί να αποφύγει η εταιρεία της ίδιας της απολύσεις. Μετά υπάρχουν ε, κάποιες προτάσεις για τα κριτήρια παρέμβασης του ταμείου πρέπει η ευρωπαϊκή πολιτική να μπορεί να γνωρίζει πώς θα προσαρμοστεί σε κάθε οικονομική κρίση. Τέλος, θέλουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, αλλά και πιο βιώσιμη αποτελεσματικότητα για τους εργαζομένους καθώς και μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των κρατών μελών της Ευρώπης. Γιατί Τελικά, να θυμόμαστε ότι τα Ταμείο προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση δεν υποκαθιστά την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων, ούτε και την κοινωνική νομοθεσία των κρατών μελών. Κάποια μπορεί να έχουν πιο αυστηρή νομοθεσία, κάποια όχι. Δεν πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των δύο. Το Ταμείο πρέπει να ενθαρρύνει εξάλλου την υιοθέτηση νομοθεσίας και εθνικής. Ευχαριστώ. Αρχίζει η συζήτηση. Ο κύριος Χέντελ. Όχι, μια στιγμή. Η κυρία Κονέλσον είχε σηκώσει προηγουμένω το χέρι τη πριν από, από τον κύριο Χέντελ. Κονέλσον και μετά Έντελ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Στην ακρόαση που κάναμε πριν από δύο-τρεις εβδομάδες ελέγξαν πάρα πολλά για τη διαδικασία του Ταμείου παγκοσμιοποίησης που αφορούσαν ε, το γεγονός ότι ορισμένα πράγματα δεν πήγαιναν πολύ καλά. Βέβαια τα κράτη-μέλη θεώρησαν θετικό ότι υπήρχε αυτό το ταμείο. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ θετικό ότι προηγήθηκε η συζήτηση για τις ε, κατευθυντήρες γραμμές για την απασχόληση και τώρα το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης, γιατί συνάπτονται τα δύο θέματα. Αν τα κράτη-μέλη πάνε σοβαρά την ε, Ευρώπη του 2020 και τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση θα προχωρήσουν στην πρόληψη της ανεργίας, θα επενδύσουν στην οικονομία μας με τέτοιο τρόπο ώστε αυτές οι μαζικές απολύσει, ιδίω σε πεπαλαιωμένους μέσα σε εισαγωγικά οικονομικούς τομεί, δεν θα γίνουν πραγματικότητα. Αλλά προς το παρόν νομίζω ότι είναι σημαντικό να υπάρχει κάποια χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις κατεπίγουσας ε, ανάγκης. Δεν ξέρω εδώ αν χρειάζεται μια χωριστή γραμμή του προπολογισμού όπως αυτή που προτείνει η κυρία Σωτιέ αν Αυτός είναι ο μόνος ή ο καλύτερος τρόπος, ίσως ο κύριος Πόρτας από την Επιτροπή Προϋπολογισμών θα μπορούσε να μας δώσει περισσότερες ιδέες γιατί γνωρίζει καλύτερα τις ε, δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν και ίσως θα ήταν απαραίτητο να έχουμε μεγαλύτερη συνεκτικότητα μεταξύ αυτής της ε, πολιτικής και άλλων πολιτικών. Το είδαμε αυτό σε προηγούμενες περιπτώσεις πέρσι. ότι η απασχόληση εξαρτάται από πολλούς άλλους τομείς πολιτικής, όπως είναι η βιομηχανική πολιτική, η πολιτική ανταγωνισμού, η πολιτική για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, περιφερειακή πολιτική, η πολιτική σε επίπεδο διεθνούς εμπορίου κτλ. Πιστεύω λοιπόν ότι η αξιολόγησή μας θα πρέπει να εστιάσει και σε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη συνοχή και συνεκτικότητα μεταξύ των διαφορετικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να λειτουργήσει καλύτερα και το Ταμείο αυτό. Απλώς λοιπόν θα ήθελα να διερευνηθούν όλες αυτές οι δυνατότητες για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε και στην Ιρλανδία όταν θα πάμε εκεί για να δούμε καλύτερα πώς λειτουργεί αυτό το ταμείο. Σας ευχαριστώ κύριος Χέντελ και κυρία Λίνκεβιτς Ιούτια. Μετά κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, για την έκθεση, <clears throat> πιστεύω καταρχήν ότι είναι μια πολύ πετυχημένη έκθεση, Έχω όμως παρόλα αυτά να κάνω κάποιες παρατηρήσεις, όπου θεωρώ ότι αυτό θα μπορούσε να βελτιώσει ακόμα περισσότερο την έκθεση στο παρελθόν το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης φάνηκε σαν ένα καλό μέσο για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα κράτη-μέλη τις ανάγκες της ε, προστασίας των εργαζομένων μετά από την ε, απόλυσή τους, αλλά εδώ έχει να κάνει και με το θέμα, έχω κάποιες, ε, κάποια ερωτηματικά, για τα συνοδευτικά μέτρα. Παραδείγματος χάρη στο σημείο 3 αναφέρεται ότι πρέπει να συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι στην διατύπωση αιτήσεων για το ε, Ταμείο Παγκοσμιοποίησης, ίσως μπορούμε να το ενισχύσουμε αυτό, να είναι δεσμευτική η ανάγκη παρουσίας τους και όχι μόνο εκ των υστέρων να γίνονται ε, διαβουλεύσεις για να υπάρχει κάποια παρουσία των κοινωνικών εταίρων. Θα πρέπει να συμμετέχουν εξ αρχής στην διατύπωση και τη διαμόρφωση της όλης διαδικασίας. Ένα δεύτερο σημείο που είναι ακόμα πιο σημαντικό για μένα <clears throat> πολλοί από εμά θυμούνται τα γεγονότα του προηγούμενου φθινοπόρου όταν η εταιρεία Dell στην Ιρλανδία ζήτησε να εφαρμοστεί το ταμείο αυτό, ζητήθηκε μια βοήθεια 15 εκατομμύρια όταν κλείσαν τα εργοστάσια της Dell που οι υπολογιστέ στην Ιρλανδία. Η εταιρεία Dell είχε σαν στόχο με το κλείσιμο αυτό των εγκαταστάσεων να πάει στην Κίνα αλλά μετά από μερικές εβδομάδες δεν μεταφέρθηκε στην Κίνα, αλλά στην Πολωνία. Καλό για την υποδομή στην Πολωνία, αλλά αυτό σήμαινε ότι υπήρξε, ε, εποφελήθηκε η εταιρεία από μια χρηματοδότηση 48 εκατομμυρίων από ένα άλλο ταμείο και στην περίπτωση αυτή πήρε κατά κάποιο τρόπο μια διπλή επιδότηση. Και μιλάμε για μια εταιρεία που πριν από στο παρελθόν μέσα σε τρία χρόνια είχε κέρδη δισεκατομμύριων. Θα ήθελα λοιπόν να σκεφτούμε καλύτερα πώς μπορούμε να αποφύγουμε τέτοιες καταχρηστικές χρησιμοποιήσεις των ευρωπαϊκών πόρων και επομένως να εξασφαλίσουμε ότι το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης θα εμπλέκεται μονάχα σε αναδιαθρώσεις που πράγματι να τεκμηριώνεται ότι είναι απαραίτητες και συγχρόνως ότι έχει σαν στόχο να αντιμετωπίσει τις πραγματικές κοινωνικο-οικονομικές ζημίες που προέρχονται από μια μεταφορά επιχείρησης, μια μετεγκατάσταση επιχείρησης. Και οι επιχειρήσεις οι ίδιες θα πρέπει και αυτές να συμβάλλουν εν μέρη στην αντιμετώπιση αυτού του κόστους. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν να το λάβει αυτό υπόψη η συγγήτρια στην εκθεσή της. Μήπως θα πρέπει να υπάρχει μια μεγαλύτερη, πιο ε, πιο δεσμευτικές προϋποθέσεις για την προσφυγή στο Ταμείο Παγκοσμιοποίησης και αυτό να αντανακλάται στην εκθεσή της. Συγγνώμη, κυρία Ευχαριστώ. Ε, να ευχαριστήσω κατά πρώτον την κυρία Σαρτιέ για τις πολύ καλές της προτάσεις και να υπογραμμίσω κάποιες ιδέες να πω ότι η χώρα μου, η Λιθουανία, έχει ζητήσει με αίτηση της βοήθεια και στήριξη από αυτό το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Διότι ο χώρος των οικοδομών, ο κατασκευαστικός τομέας, ο τομέας ε, της κατασκευής ρούχων, Όλα αυτά επηρεάστηκαν από την κρίση. Χρειάστηκε λοιπόν η Λιθουανία την συνδρομή του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και αυτή ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη. Θυμίζω το σημείο που έθεσε ένας συνάδελφος που ρωτούσε εάν υπάρχει τρόπος να διοργανωθούν διαβουλεύσεις της δικής μου χώρας και της δικής του συγκεκριμένα ενδιαφερόταν να μάθει κατά πόσον ήταν δυνατή η ανταλλαγή καλών πρακτικών. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Αναφέρεται και στο σημείο 4 ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθούν επαφέ μεταξύ των κρατών μελών, να ανταλλάσσονται καλέ πρακτικέ, διότι ακόμη κάποια από τα κρατημέλη δεν ε, είχαν προσφύγει στο Ταμείο για στήριξη. Ίσως γιατί δεν το γνώριζαν, ίσως γιατί δεν υπήρξε η ανάγκη. Ε, Στη Λιθουανία είχα αρκετέ φορέ την ευκαιρία να συζητήσω με εργαζομένου αρκετών επιχειρήσεων και όλοι μου τόνισαν ένα πρόβλημα σημαντικό που και εσεί το αναφέρατε. Όταν μιλάμε για μια χρονική περίοδο 1,5 έτους, αυτή η περίοδος είναι ιδιαίτερα παρατεταμένη για να ε, κανείς, για να περιμένει κανείς να ωφεληθεί από το Ταμείο. Όταν κάποιος απολύεται χρειάζεται άμεσα βοήθεια όταν οι απολύσει είναι μαζικέ. Στο σημείο 2 λοιπόν, εκεί που μιλάτε για την απλούστευση των διαδικασιών, για την μείωση των προθεσμιών εξέταση των αιτήσεων. Αυτό δείτε το. Δείτε το γιατί διαφορετικά ο κόσμος δεν θα μας εμπιστεύεται πλέον, δεν θα εμπιστεύεται την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα λέει ότι είμαστε μόνο γραφειοκράτες και τεχνοκράτες που παράγουμε τόνους επιτόνων χαρτιού. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο στηρίζω την ιδέα σας να διατηρηθεί το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση που είναι και αναγκαίο αλλά να εργάζεται πολύ πιο γρήγορα. Ευχαριστούμε κυρία Φιγκέιρα εδώ. Ευχαριστώ. Έχουμε εργαστεί αρκετά στην ομάδα εργασίας που ασχολείται με το θέμα αυτό επί της ουσίας, με το θέμα της, ε, του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν διάφορα προβλήματα, που και εδώ ακούστηκαν κάποιες επιλογές, ακούστηκαν όπως η περίπτωση της ΔΕΛ και άλλες παρόμοιες. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε κατά πόσον μπορούμε να βελτιώσουμε την κινητοποίηση αυτού του ταμείου και από διαφορετικές προοπτικές. Όμως αυτή τη χρονική συγκυρία, αυτό που μας απασχολεί κατά κύριο λόγο, είναι η συγχρηματοδότηση. Χώρες οι οποίες έχουν σοβαρά προβλήματα δημοσιονομικά και δεν προσφεύγουν στο ταμείο, δεν έχουν δυνατότητα 35% συγχρηματοδότησης, υποχρεωτικής συγχρηματοδότησης ακόμη και μετά την αναθεώρηση των προγραμμάτων. Γι' αυτόν τον λόγο προκύπτουν επίσης από χώρες με καλύτερες δημοσιονομικές συνθήκες και δεν υπάρχουν αιτήσει από χώρες με σοβαρότατα προβλήματα ανεργίας αλλά και σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα. Άρα το πρόβλημα αυτό θα πρέπει σοβαρά να το σκεφτούμε στην περίπτωση μεταρρύθμισης του Ταμείου αυτό το σημείο είναι κεντρική σημασία. Θα πρέπει να το εξετάσουμε και να θέσουμε εδώ κάποια πρόταση σχετικά. Να υποβάλουμε κάποια πρόταση γιατί κάτι τέτοιο είχαμε κάνει και κατά τη στιγμή της ίδρυσης του Ταμείου. Τότε που μιλούσαμε για 80% κοινοτικής χρηματοδότησης και 20% εθνικής χρηματοδότησης. Στην αρχή λοιπόν μείναμε στο 50% από κάθε πλευρά και έπειτα η Επιτροπή αναθεώρησε προσωρινά στο 65% το ποσοστό αυτό. Όμως νομίζω ότι μια ουσιαστική μεταρρύθμιση του Ταμείου θα πρέπει να λάβει υπόψη και αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι καθοριστικής σημασίας πέραν άλλων σημαντικών που ούτω ή άλλω αναφέρθηκαν και με, με τις οποίες συμφωνώ. Καλύτερη ενημέρωση, διάδοση των καλών πρακτικών, το πρόβλημα της απαγόρευσης μετατόπισης και μετακίνησης των πολυεθνικών επιχειρήσεων και προφανώς Υπάρχουν επιχειρήσεις που δεν έχουν ανάγκη να κάνουν κάτι τέτοιο και απλώς κοιτάζουν να αυξήσουν τα κέρδη τους. Υπάρχουν και άλλα σημεία στα οποία θεωρώ ότι επιδέχεται το κείμενο βελτίωσης, όμως αυτές είναι γενικές κατευθύνσεις που θα πρέπει να ακολουθήσει η συζήτησή μας και συμφωνώ με τους περισσότερους από του συναδέλφους που τοποθετήθηκαν. Ευχαριστώ. Κυρία Βέβαια, υπάρχουν ε, οι τεχνικοί του προϋπολογισμού που γνωρίζουν περισσότερο για τα οικονομικά, για τη διαδικασία του προϋπολογισμού. Επομένως θα ήθελα εγώ να θέσω το ερώτημα αυτό της ε, μονιμότητος της γραμμής του προϋπολογισμού. Είναι ένα ερώτημα που ήθελα να θέσω προς την Κομισιόν, αν θεωρεί ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο από τεχνική άποψη. Εγώ πιστεύω ότι λείπει μια νομική βάση καταρχήν και αυτό είναι ένα ερώτημα του αν μπορούμε να έχουμε μια νομική βάση την οποία θα χρησιμοποιήσουμε και από πολιτική άποψη Όποιο ξέρει πώς λειτουργούν οι διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο, ξέρει ότι είναι πολύ περιορισμένε οι δυνατότητε να λειτουργήσει αυτό το Ταμείο. Πολλέ φορέ στο παρελθόν έχουμε χρησιμοποιήσει για του σκοπού αυτού το, το αποθεματικό, το ειδικό αποθεματικό. Υπάρχει όμω μια δυνατότητα να δούμε αν μπορούμε να φτιάξουμε κάποιο σύστημα μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι εμείς ως Κοινοβούλιο έχουμε τη δυνατότητα συναπόφασης μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και αντίθετα με τα θέματα της, των, προ, δημοσιονομικών προοπτικών έχουμε μια μεγαλύτερη δυνατότητα επιρροής χάρη στη Συνθήκη της Λισαβόνας ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Γι' αυτό, βάσει της εμπειρίας που έχω με τα διαφορετικά ταμεία, νομίζω ότι θα έχουμε περισσότερες δυνατότητε στα πλαίσια του κοινωνικού ταμείου. Ελπίζω λοιπόν ότι αυτό θα μπορέσει να γίνει πραγματικότητα. Μπορούμε να τονίσουμε στα κράτη-μέλη ότι αυτό τους δίνει και μεγαλύτερη ευελιξία, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε αν θα πρέπει να δώσουμε τόσες πολλές δυνατότητες στα κράτη-μέλη σε βάρος της ευρωπαϊκής ε, ε, αντιμετώπισης. Είναι λιγότερο λοιπόν ε, ιδανικό αυτό και ευνοϊκό από το παρουσίασε ο κύριος Μπαρόσο, αλλά ενδεχομένω να είναι πιο πραγματιστική αυτή η αντιμετώπιση μέσω του κοινωνικού ταμείου. <clears throat> Γιατί βλέπουμε ότι η διαδικασία κινητοποίηση του αποθεματικού στον προπολογισμό απαιτεί χρόνο και πολλή προσπάθεια και πιστεύω ότι με το με τη χρήση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, με τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου μπορούμε να έχουμε και την ευελιξία που απαιτείται και την ικανότητα ταχύτερη κινητοποίηση αυτού του εργαλείου. Θα έπρεπε λοιπόν ίσω ενδεχομένω να σκεφτούμε περισσότερο και εναπόκειται <clears throat> βέβαια στους ειδήμονε του προπολογισμού να την κάνουν πιο λειτουργική και στην εισηγήτρια. Θα ήθελα να έχω και την απόψη Κομισιόν σχετικά. Ευχαριστώ. Κυρία εισηγήτρια, προφανώ θα έχετε πολλέ τροπολογίε από την κυρία Σρέντερ και επομένως μια καλή βάση διαπραγματεύσεων. Προτού δώσω το λόγο στον Διευθυντή του Ταμείου που είναι παρόν μεταξύ μας για αυτό το συγκεκριμένο θέμα του προϋπολογισμού, επειδή ακριβώς του ετέθη αυτό το ερώτημα, θα ήθελα να τονίσω τρία σημεία τα οποία βρίσκονται στην έκθεσή σας και τα οποία έχουν μεγάλη σημασία. Πέραν τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και του κοινωνικού διαλόγου που πιστεύω ότι πρέπει να τονιστεί και πάλι. Είδαμε την συγκεκριμένη περίπτωση της ΔΕΛ, η οποία είναι παραδειγματική, σαν αντιπαράδειγμα κατάστασης που δεν πρέπει να επαναληφθεί στο μέλλον και όπου φάνηκε ότι η έλλειψη κοινωνικού διαλόγου υποβάθμισε την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της ε, παρέμβασης της ευρωπαϊκή Ένωσης και της διαδικασίας. Ένα δεύτερο στοιχείο, κυρία Συγήτρια, δεν θα σας εκπλήξω, είναι το θέμα της συνεκτικότητας των πολιτικών της Κομισιόν. Πέραν της δικής μας εστίασης σε σχέση με τη λειτουργία του Ταμείου αυτού, <clears throat> θα πρέπει η Κομισιόν να δράσει σαν ένα συλλογικό όργανο και όχι σαν απλό ασυνάρτητο άθροισμα γενικών διευθύνσεων ή επιτρόπων που δεν γνωρίζει η δεξιά του τι πει η αριστερά του ή ο δεξιό επίτροπο τι κάνει ο αριστερό επίτροπο. Θα χρειάζεται λοιπόν μια μεγαλύτερη συνεκτικότητα στι δράσει τη Κομισιόν. Και το τρίτο σημείο είναι το θέμα τη ανισότητα πρόσβαση των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τη χρησιμοποίηση του Ταμείου. Εδώ δεν είναι ριζοσπαστικό αυτό το οποίο προτείνουμε. Γιατί στην περίπτωση της Λιθουανίας έχουμε πράγματι σημαντική χρησιμοποίηση του Ταμείου. Γνωρίζουμε όμως ότι για τα κράτη-μέλη η δυνατότητά τους προσφυγής σε αυτό το Ταμείο είναι ποικίλουσα. Και για τους στόχους του Ταμείου αυτού, που είναι στόχοι που αφορούν τις ανάγκες των εργαζομένων και όχι την κατάσταση της ίδιας αυτής της χώρας η οποία πρέπει να συγχρηματοδοτήσει, προκύπτει μια δυσκολία η οποία τη στιγμή αυτή που έχουμε να αναθεωρήσουμε τη λειτουργία του ταμείου αυτού θα μπορούσε να εξεταστεί πολύ πιο προσεκτικά. Ξέρω ότι τροποποιήθηκε πρόσφατα ο κανονισμός του Ταμείου προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση, αλλά αυτή είναι ίσως μια <clears throat> βελτίωση που γίνεται ενώ βρισκόμαστε εν πορεία και ίσως η έκθεση την οποία εκπονείτε εσείς μαζί με τον Μιγγέλ Πόρτος, στον οποίο θα δώσω το λόγο, ίσως η έκθεσή σας θα μπορέσει να εξετάσει αν είμαστε στις βέλτιστες συνθήκες χρησιμοποίησης αυτού του Ταμείου. Κύριε Πόρτας, τώρα ή μετά από τον εκπρόσωπο του Ταμείου. Σας δίνω το λόγο λοιπόν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι συντομότατος. Υπάρχει ένα σύνολο προτάσεων και συστάσεων που διατυπώθηκαν από την κυρία Σατιέ και αυτές προκύπτουν και από τις συζητήσεις που έλαβαν χώρα στις δύο επιτροπές μας, απασχόλησης και προϋπολογισμών θα έλεγα, ότι σε γενικές γραμμές αντανακλώνται ή πρέπει να αντανακλώνται και στην τελική έκθεση η οποία θα προκύψει και η οποία θα έρθει σε ψηφοφορία. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν την κυρία Σόρτιε για την πολύ καλή βάση εργασίας που δημιουργήσε. Και τώρα θέλω να σταθώ μονάχα σε τρία σημεία τα οποία αναφέρθηκαν και να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Ετέθη το ερώτημα του αν η καλύτερη λύση θα ήταν να ενσωματώσουμε στον προϋπολογισμό το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, δηλαδή να είναι ένα ταμείο το οποίο περιλαμβάνεται στον προπολογισμό. Κάτι να άποψή μου αυτό είναι η καλύτερη λύση εν του μέλλοντο. Αλλά συμφωνώ με την παρατήρηση η οποία έγινε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν οι πολιτικές προϋποθέσεις, ιδίως σε επίπεδο Συμβουλίου, ώστε να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι η πρόταση επί τη βάση τη οποία θα πρέπει να προχωρήσουμε είναι να υπάρξει μια σημαντική απλοποίηση των διαδικασιών στο τωρινό, πλαίσιο, το τωρινό νομικό πλαίσιο μέχρι το 2013 και επέκεινα το 2013 να υπάρξει μια στεναρή θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να εξασφαλίσουμε ότι το Ταμείο αυτό προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση θα μπορέσει να είναι ένα φυσιολογικό ταμείο με τη δική του χρηματοδότηση από το 2013 που θα ισχύσουν οι επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Αυτό είναι μια πολιτική μάχη που θα πρέπει να δώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα πρέπει να δώσουμε τα σωστά πολιτικά μηνύματα σε ό,τι αφορά κάτι που είναι ένα από τα μεγαλύτερα πολιτικά προβλήματα, κοινωνικά προβλήματα, συγγνώμη, που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, που είναι η αύξηση των απολύσεων μέσα από τις συλλογικές απολύσεις. Επίσης, Συμφωνώ με πολλές από τις προτάσεις οι οποίες διατυπώθηκαν είτε σε ό,τι αφορά τη συγχρηματοδότηση, το πρόβλημα λοιπόν της συγχρηματοδότησης και της διαφοράς μεταξύ των πλουσίων περιοχών και των φτωχότερων περιοχών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης σε σχέση με το να είναι δεσμευτική, υποχρεωτική δηλαδή η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων κάθε φορά που υπάρχει μια κατάσταση ε, που προβλέπει συλλογικές απολύσεις. Υπάρχει άλλο ένα ερώτημα, όπου μάλλον θέλω να θέσω ένα ερώτημα και όχι μια απάντηση. Ήταν το ερώτημα που έθεσε ο συνάδελφος Χάντεο. Πώς, Χάντελ, πώς λύνονται προβλήματα όπως αυτό της εταιρείας Dell. Αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό θέμα και στην Επιτροπή Απασχόλησης και στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Ουσιαστικά είμαστε όλοι τα θύματα μιας παγίδας στην οποία πέσαμε. Δηλαδή η επιχείρηση αυτή μπορεί να κάνει τις συλλογικέ απολύσεις. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε μην το κάνετε αυτό. Υπήρξαν εργαζόμενοι οι οποίοι απολύθηκαν σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακόμα και αν αυτή η απόλυση ήταν αποτέλεσμα μιας μετεγκατάστασης της επιχείρησης αυτής μέσα στην ίδια την εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ερώτημα είναι, μπορούμε εμείς από πολιτική έποψη να πούμε ότι αυτό το ταμείο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτούς οι οποίοι κάνουν μετεγκατάσταση μέσα στην εσωτερική αγορά. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Δεν μπορούμε αυτό να το θέσουμε σαν προϋπόθεση. Εμείς ίσως χρειαζόμαστε μια διαφορετική έκθεση η οποία να προβλέπει τις προϋποθέσεις και το τίμημα μιας μετεγκατάστασης πολυεθνικών εταιριών μέσα στην εσωτερική αγορά. Θα πρέπει λοιπόν να αποφασίσουμε ποιο είναι το τίμημα το οποίο πρέπει να καταβάλει μια πολυεθνική εταιρεία σε περίπτωση συλλογικών απολύσεων εν ώψη με την κατάσταση στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν σαν στόχο μονάχα την αύξηση των κερδών. Φυσικά δεν πρέπει σε αυτή την περίπτωση να πληρώσουν την ύφη οι απολυόμενοι εργαζόμενοι. Αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι μέσα σε αυτή την έκθεση δεν είμαι σε θέση να δώσω μια λύση σε αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον διευθυντή του Ταμείου, τον κύριο Γιώργενσεν, και μετά το λόγο και πάλι στην εισηγήτριά μας. Κύριε Γιώργενσεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστούμε και για την έκθεσή σας που την μελετήσαμε, συμπεριλαμβάνει ορισμένα πολύ χρήσιμα και διευκρινιστικά στοιχεία που από ό,τι βλέπω μέχρι στιγμής δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να τα δεχτούμε. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι είναι σημαντικό να πούμε ότι οι εταιρείε δεν λαμβάνουν χρηματοδότηση από το Ταμείο. Η Dell δεν έλαβε χρηματοδότηση από το Ταμείο ούτε στην Ιρλανδία ούτε και αλλού. Οι απολυμμένοι εργαζόμενοι της Dell στηρίχθηκαν και στηρίζονται όμως από μέτρα από το Ταμείο. Δεύτερον, στην περίπτωση της Dell δεν είχαμε εσωτερική επανεγκατάσταση εντός της εσωτερικής αγοράς. Υπήρχε συγκεκριμένη διαφορά μεταξύ του τι παραγόταν στην Ιρλανδία και το τι παραγόταν στην Πολωνία. Δεν υπήρξε δηλαδή μεταφορά των παραγωγικών δυνατοτήτων εντός της εσωτερικής αγοράς. Τώρα, όσον αφορά τον προϋπολογισμό. Η ιδέα να υπάρξει συγκεκριμένη γραμμή για το Ταμείο εντός των επόμενων δημοσιονομικών προοπτικών είναι κάτι που συζητάμε αυτή τη στιγμή γιατί προφανώς δεν μπορεί να εισαχθεί, να εισαχθεί τώρα συγκεκριμένη γραμμή για το Ταμείο στις υπάρχουσες δημοσιονομικές προοπτικές και δεν θα μπορούσαμε να, να δημιουργήσουμε και νομοθεσία αυτή τη στιγμή τώρα. Άρα, η ιδέα που αναφέρει και η συγγήτρια είναι για τις επόμενες δημοσιονομικές πρόπτικες το Ταμείο Αντιμετώπισης της Παγκοσμιοποίησης όπως και τα υπόλοιπα ταμεία θα έπρεπε να έχει τα διδική του γραμμή στον προϋπολογισμό. Και στο Γκέτεμπορκ ο Επίτροπος ανέφερε ότι σκέφτεται να κάνει πρόταση για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Βεβαίως αυτό θα πρέπει να τύχει πολιτική συζήτηση εντός της Κομισιόν και των δημοσιονομικών αρχών Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε εμείς τώρα. Αυτό που είπε και ο κύριος Πόρτας να συνεχίσουμε να απλοποιούμε και να κάνουμε πιο αποτελεσματικές τις διαδικασίες. Αυτό ήδη το έχουμε κάνει εσωτερικά στην Κομισιόν, όπου συγχωνεύσαμε δύο διαδικασίες σε μία και κερδίσαμε κατά μέσο όρο 22 ημέρες, το χρόνο που χρειαζόμαστε κάθε φορά. Και τώρα εξετάζουμε το νέο βήμα το επόμενο βήμα στην απλοποίηση που αφορά την λήψη αποφάσεων για τη χρηματοδότηση και την πληρωμή των κρατών μελών. Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε περίπου 55 ημέρες για την πληρωμή από τη στιγμή που υπάρχει συμφωνία της Δημοσιονομικής Αρχής. Νομίζουμε ότι βρήκαμε τρόπο να μειώσουμε αυτό τον χρόνο στις 14 ημέρες, δύο εβδομάδες δηλαδή. Κερδίζουμε ένα χρόνο και, ένα μήνα με συγχωρείτε ή και περισσότερο. Επίσης, προσπαθούμε να βρούμε τρόπους που θα μας επιτρέψουν να απλοποιήσουμε τη διαδικασία διερεύνησης του φακέλου. Ενδεχομένως θα μπορούσαμε να εργαζόμαστε σε περισσότερες γλώσσες ώστε να μην χρειαζόμαστε τόσες πολλές μεταφράσεις. Βεβαίως, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα τεχνικά βήματα τα οποία απαιτούνται εξαιτίας της ειδική κατάστασης που ισχύει όσον αφορά τον προϋπολογισμό του Ταμείου. Να πω επίσης ότι όλες οι αποφάσεις του Ταμείου λαμβάνονται από το Κολέγιο των Επιτρόπων από την Επιτροπή ως συλλογικό όργανο. Όλα λοιπόν τα μέλη της Επιτροπής μπορούν να εξετάσουν κάθε μία υπόθεση και να διασφαλίσουν ότι κάθε μία αίτηση συμβαδίζει με τις πολιτικές του χαρτοφυλακίου τους. Άρα υπάρχει διαβούλευση εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν ληφθεί η απόφαση και η απόφαση λαμβάνεται από το σύνολο των επιτρόπων σε κάθε περίπτωση. Κάτι ακόμη που θα ήθελα να τονίσω που ανέφερε η εισηγήτρια όσον αφορά την ευελιξία των κριτηρίων παρέμβασης. Ειδικά όταν πρόκειται για διασυνοριακές ε, αιτήσει οι αιτήσει πολλών κρατών μελών. Στο σημείο 9 αναφέρεται ότι ίσως θα μπορούσαν να επεκταθεί η περίοδος αναφοράς και οι παράμετροι. Κοιτάξτε, η περίοδος αναφοράς αναφέρεται στον κανονισμό και όλοι οι παράμετροι, όλες οι παράμετροι που αφορούν το μέγεθος και τα λοιπά επίσης αναφέρονται στον κανονισμό. Αυτά τα θέματα λοιπόν μπορούμε να τα εξετάσουμε όταν υπάρξει αναθεώρηση του κανονισμού, αλλά όχι υπό άλλες συνθήκες. Και περνάω στο ένα τελευταίο σημείο. Είναι προφανές ότι ο παρόν κανονισμός με τις τροποποιήσεις που έγιναν πέρυσι, λίγη τέλη 2011. Άρα θα έχουμε μία μεταβατική περίοδο το 2011 όπου θα μπορούσαμε να αποφασίσουμε αν θέλουμε να σταματήσουν οι παρεκκλήσεις που ισχύουν ή αν θέλουμε να τις παρατείνουμε εξαιτία της συνέχισης της οικονομικής κρίσης. Όμως αυτό έχει να κάνει και με την πολιτική απόφαση για το κατά πόσο θα θέλαμε περαιτέρω συντονισμό του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση με τα διαρθρωτικά ταμεία. Όμως δεν μπορώ να σας απαντήσω σήμερα σε αυτό το ερώτημα, ούτε είναι και δική μου αρμοδιότητα. Σας ευχαριστούμε όμως σε κάθε περίπτωση η συζήτηση αυτή θα θα διευκολύνει και την λήψη απόφαση από το Κοινοβούλιο. Είσαι Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που παρενέβησαν και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου για τις προτάσεις αυτές που μας υποβάλλονται. Βεβαίως στην Επιτροπή των Προϋπολογισμών θα αφήσω την ευθύνη για την συγκεκριμένη ανάλυση των προτάσεων και την δημοσιονομική μας διοργάνωση. Όμως πολύ σωστά διακριβώνεται εδώ ότι με το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο θα αρχίσει να ισχύει και η συγκεκριμένη πρόταση. Για την επιχείρηση Dell όλοι στην ομάδα εργασίας παρακολουθήσαμε την περίπτωση της επιχείρησης αυτής και την λήψη των αποφάσεων από το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Οι αποφάσεις αυτές αφορούσαν αποκλειστικά και μόνον το πώς θα ωφεληθούν οι εργαζόμενοι και μια μικρή προσθήκη σε όσα υπόθησαν ότι κατά την υλοποίηση, το άνοιγμα μάλλον ως εργοστασίου στην Πολωνία, σκοπός ήταν να παράγονται προϊόντα τα οποία ήταν ιδιαίτερα σημαντικά για αυτήν την αγορά, για φορητούς υπολογιστές πρώτο. αγορά που βρισκόταν σε ε, αύξηση σε εκείνη την ε, περιοχή. Ενώ στην Ιρλανδία παραγόνταν υπολογιστέ γραφείου, desktop, οι οποίοι ούτω ή άλλω ήταν μια αγορά που βρισκόταν σε συρρήκνωση. Αυτό λοιπόν ω προ τον, ως προσανατολισμό της επιχείρησης σκοπό δεν είχε να πλήξει την παραγωγή στην Ιρλανδία. Η μετακίνηση αυτή έγινε για την παραγωγή μια σειράς νέων προϊόντων. Και όπως είπε και η κυρία Κορνέλισεν, μια μικρή κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία αποτελούμενη κατεξοχήν από μέλη της ομάδας εργασίας ε, για το Ταμείο Προσαρμόγης στην Παγκοσμιοποίηση. Θα πάμε στην Ιρλανδία αυτή και όλα στην εβδομάδα στην ΔΕΛ, για να δούμε τι έγινε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο. Οφελήθηκαν οι εργαζόμενοι ή όχι. Η επαγγελματική του ενσωμάτωση επιδιώχθη ή όχι και θα μπορέσουμε να μιλήσουμε και με επικεφαλής επιχειρήσεων, υπευθύνου του εργοστασίου, αλλά και τους εκπροσώπους κατεξοχήν των εργαζομένων. Να προσθέσω επίσης ότι ακόμη και για τα πρώτα κονδύλια που δόθηκαν από το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, μετά από εξακρίβωση υπήρξαν και κάποιες επιστροφές, καθόλου αμελητές, οι οποίες απαιτήθησαν κιόλας, διότι η χρήση δεν ήταν η αρμόζουσα. σημειώνω την αίτηση για ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ κρατών μελών, όπως πολύ σωστά το επεσήμανε μία συνάδελφος. Σημείωσα επίσης την παρέμβαση της κυρίας Φιγκεϊρέδου για την εθνική συγχρηματοδότηση και τα ποσοστά τα υποχρεωτικά όπως αναθεωρήθηκαν μετά το έργο του Κοινοβουλίου, βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει πεδίο ε, ελεύθερο για να εργαστούμε, για να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητά μας. Έπειτα, αυτό που έρχεται κατόπιν είναι ότι θέλουμε να αναπτυχθεί ο κοινωνικός διάλογος, θέλουμε εντός των επιχειρήσεων και καθόλου τη διάρκεια της διαδικασίας να υπάρχει συζήτηση. Εδώ και για την ΤΕΛ και για άλλους. Θα πρέπει να είμαστε πολύ περισσότερο απαιτητικοί κατά την εξέταση των θεμάτων μας. Στο σημείο αυτό, λοιπόν, είμαι ιδιαίτερα δραστήρια και εγώ ίδια. Δεδομένων των παρατηρήσεων που έγιναν, προσυπογράφω σε πάρα πολλές από τις παρατηρήσεις που ακούστηκαν και θα φροντίσω τις επόμενες ημέρες να έρθω σε επαφή με τους διάφορους συναδέλφους για να δούμε κατά πόσον μπορούμε να ενσωματώσουμε, να ενδυναμώσουμε τη μια ή την άλλη γραμμή της έκθεσης που σε κάθε περίπτωση συντάχθηκε πλήρη ευσυνειδησία. Σας διαβεβαιώ ότι είμαι στη διάθεσή σας γιατί έχουμε τουλάχιστον μια εβδομάδα ακόμη μπροστά μας για να φροντίσουμε να κάνουμε τις απαραίτητες συμπληρώσεις που θα κάνουν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό το σχέδιο αυτογνωμοδότηση. Διότι για την αποτελεσματικότητα τη Ευρώπη εργαζόμαστε και για το όφελο των εργαζομένων. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια. 8 Ιουνίου στις 12 η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. 23 Ιουνίου η συζήτηση. 24 ψηφίζουμε στην Επιτροπή μας. Η Επιτροπή Προπολογισμών με την οποία αποφασίζουμε από κοινού θα αποφανθεί στις 14 Ιουλίου. Έχουμε ολοκληρώσει λοιπόν και με το σημείο αυτό στην ημερήσια διάταξη και ερχόμαστε τώρα στο σημείο 14. Πριν αυτού, να σας ενημερώσω ότι προς την συνάδελφο την κυρία Γιασλοβιέτκα, η οποία έπαθε καρδιακή προσβολή κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης της αντιπροσωπείας μας στην Κίνα, έστειλε λοιπόν μήνυμα που εκφράζω την ελληνική εκ μέρους όλων μας για ταχεία ανάρρωση από μέρους μας. Είναι σημαντικό νομίζω συνάδελφοι να το γνωρίζετε και εσείς ότι επιστάλλει αυτό το μήνυμα μπορεί να χρειαστεί και εσείς να αναλάβετε δράση προσωπικά. Στο σημείο 14 λοιπόν, η θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο προπολογισμού του 2011 όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο του Ματρία, Επιτροπή. Το σημείο αυτό προβλέπει να σας παρουσιάσω το σχέδιο γνωμοδότησης που θα επιβάλλουμε. Το πλαίσιο εντό του οποίου εξετάζουμε το σχέδιο γνωμοδότηση τώρα. Να σα το θυμίσω διότι δεδομένων των προηγούμενων διαδικασιών τα πράγματα έχουν αλλάξει αρκετά με τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνα. Και ιδίω γιατί η διαδικασία εφεξής γίνεται με μία και μόνη ανάγνωση και με τη θέσπιση Επιτροπής Συνδιαλλαγής για να επιτευχθεί συμφωνία. Αυτό μας επιβάλλει κατά τον ορισμό των προτεραιοτήτων μας να είμαστε ιδιαίτερα προχωρημένοι. Γι' αυτό και οι συγητές μας φρόντισαν να εντοπίσουν τις πέντε προτεραιότητες που θα υποβάλουμε για τον προπολογισμό του 2011 και να τις θυμίσω. Κατά πολέμηση της ανεργίας των νέων, εκπαίδευση των εργαζομένων, εκπαίδευση μάλλον των ανέργων, υλοποίηση τη συμφωνία με το Συμβούλιο και το, την Επιτροπή για την υλοποίηση του προγράμματος Progress, συνεργασία με τις κοινωνικές διεθνεί οργανώσεις και εργασία για καλύτερη προώθηση του θέματος της ισότητας των δύο φύλων στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν δούμε τις, ε, τους προσανατολισμούς τους οποίους έδωσε προτεραιότητα η Επιτροπή στο σχέδιο προπολογισμού του, σημειώνουμε κάποια σημεία που μας αφορούν και εμάς εμέσως. Και η στήριξη για την οικονομική ανάκαμψη και οι επενδύσεις στην νεολαία και η ανάπτυξη υποδομών για το αύριο. Σε αυτό λοιπόν το γενικότερο σκηνικό και σύμφωνα με την άποψη των εισηγητών, αποφασίσαμε για φέτος να στηρίξουμε την ε, εισαγωγή δύο πιλωτικών προγραμμάτων, νέων πιλωτικών προγραμμάτων, που θα συμπεριληφθούν στις πρωτοβουλίες ΦΑΡ που υποβαλεί η Επιτροπή. Τα δύο αυτά πολιτικά προγράμματα σχετίζονται ταυτόχρονα με αυτό που σε ωραία γαλλικά ονομάζεται Your First Real Jobs, οι πρώτε σα πραγματικέ δουλειέ, κινητοποίηση των νέων για να βρουν ε, μια θέση εργασία. Δεύτερο πιλωτικό πρόγραμμα, στήριξη τη υγεία, τη ευημερία και τη ασφάλεια στον εργασιακό χώρο των εργαζομένων ε, προχωρημένη ηλικία. Πέραν αυτών των δύο νέων πιλωτικών προγραμμάτων, προτείνουμε και εισαγωγή του συνόλου των παλιών προγραμμάτων, όπως είχαν ε, καταρτιστεί κατά τη διάρκεια των ετών και όπως τα έχει επεξεργαστεί η Επιτροπή μας. Στο σύνολο λοιπόν της νομοδότησης τρία σημεία πρέπει να εντοπίσω, σε τρία σημεία πρέπει να σταθώ, τα οποία θεωρώ σημαντικά και όπου ελπίζω ότι θα αποφανθεί και θα συμφωνήσει με τη στάση μου η Επιτροπή, ε, η δική μας Επιτροπή, για τα 100.000 ευρώ που προβλέπονται στη δημοσιονομική γραμμή για τι πληρωμέ του Ταμείου Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση, εκφράζουμε την ικανοποίησή μα. Σοβαρή αλλαγή των ε, πληρωμών από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Επαγγελματική Κατάρτιση και Εκπαίδευση, σημαντική πρικοδότηση και εδώ για το στόχο τη στρατηγική το 2020 δεν είμαστε τόσο ευχαριστημένοι και επίσης απογοήτευση για τη τέλμα στο οποίο έχουν περιέλθει δημοσιονομικές γραμμές για την οικονομική ανάπτυξη και ε, τα μέτρα κοινωνική αντιμετώπιση των μαζικών απολύσεων. Όλα όσα επηρεάζουν την ποιότητα του κοινωνικού διαλόγου χρήζουν βελτίωσης διότι αυτό είναι ένα όπλο που διαθέτουμε. Είναι η ουσία και το πνεύμα του κοινωνικού μας μοντέλου, το οποίο νομίζω περισσότερες ομάδες, εδώ οι πολιτικές ομάδες, στηρίζουν. Ιδού συνάδελφες, όσο σας προτείνω και σας θυμίζω εφόσον πρόκειται και για την πρώτη ανάγνωση, πρώτη εξέταση μάλλον του σχεδίου προπολογισμού βάσει τη συνθήκη τη Λισαβόνα, εδώ είχαμε πάρα πολλέ επαφέ ούτω ή άλλω εκ των προτέρων. Με τη συνέργεια και τη συμφωνία φυσικά, για να μην λέω συνενοχή μόνο, με τη συνεργασία λοιπόν των συγητών, για να ορίσουμε κάποιε προτεραιότητε στι συζητήσει μα με την Επιτροπή και να εντοπίσουμε τα πιλωτικά προγράμματα που θα ευνοήσουμε. Έτσι είχαμε και μια πρώτη ανταλλαγή επιστολών εξ ονόματος όλων των συναδέλφων εδώ, μια επιστολή που απευθύναμε στην κυρία Γετζε, δύσκολο, Γεντρε, Γετζεντρεύσκα, η οποία είναι επί της ουσίας εισηγήτρια στην Επιτροπή Προπολογισμών, γράμμα το οποίο όλοι νομίζω λάβατε σε αντίγραφο και που ορίζονται με τη συμφωνία των εισηγητών, οι βασικέ μας προτεραιότητες. Ιδού τα όσα ήθελα να σας πω και με μεγάλη μου χαρά να ακούσω τις αντιδράσεις σας, τι, να δεχτώ τις συνεισφορές σας για όλο αυτό το θέμα. Κύριο Θέρκαθ, συντομότατα κυρία Πρόεδρε, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι το κυριότερο σημείο που είχαμε δει με τους συντονιστές τα κυριότερα σημεία που είχαμε συζητήσει μάλλον στη συνεδρία των συντονιστών είχαν, έχουν ληφθεί υπόψη. Έχουμε την ανάγκη να μάθουμε πώς τρέχουμε με τη νέα συνθήκη της Λισαβόνας με ένα ενεργητικό τρόπο και η γνωμοδότησή μας αυτή, η πρώτη γνωμοδότηση σε αυτό το πλαίσιο κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει λοιπόν να υλοποιήσουμε όλες αυτές τις συμφωνίες που έχουμε συνάψει ως συντονιστές στο παρελθόν. Άλλοι παρεμβαίνοντες. Κυρία Λαμπέρο, όχι, δεν θέλετε. Συμφωνείτε όλοι. Είναι περιεκτικότατη αυτή η διαδικασία από τα γενοφάσκια τη. Επομένως, ίσως δεν χρειάζεται περισσότερη συζήτηση. Μονάχα μία soft διαδικασία, όπως έλεγε και ο Σακεσπύρος. από την Κομισιόν, λοιπόν, θέλετε να πείτε κάτι για τα πιλωτικά σχέδια, δεν έχετε κάποιε δυσκολίε. Κάποιο σχόλιο από την Κομισιόν έχετε το λόγο σχετικός για την Κομισιόν απλώς ευχαριστίες για το σχέδιο γνωμοδότησής σας και προφανώς η Κομισιόν υποστηρίζει τα δύο πιλωτικά σχέδια τα οποία έχουν προταθεί. Θέλω απλώς να προσθέσω σε σχέση με τα θέματα του κοινωνικού διαλόγου και εμεί συμμεριζόμαστε την ε, μνά σας και τις ανησυχίες σας για την τελμάτωση αυτής της διαδικασίας είναι προϊόν κατά κάποιο τρόπο συγκρούσεως μεταξύ γραμμών του προϋπολογισμού σε σχέση με τη χρηματοδότηση. Ελπίζουμε θα μπορέσει να επιληθεί το θέμα αυτό στο μέλλον. Ώστε να μπορέσει λοιπόν να χρηματοδοτηθεί αυτή η γραμμή η οποία υποστηρίζει τον κοινωνικό διάλογο. Το Κοινοβούλιο λοιπόν θέλει να ενισχυθεί αυτή η γραμμή του προϋπολογισμού. Κυρία Μπαστός, για το θέμα του προϋπολογισμού θέλετε να παρέμβετε ως σκιώδης. Εντάξει, τελειώνει η συζήτηση τότε. Και πρέπει να, να θεσπίσουμε προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών <clears throat> μέχρι τις 29 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι, στη συνέχεια θα εξετάσουμε στις 14 Ιουλίου τις τροπολογίες και στις 13 Σεπτεμβρίου θα γίνει η επίσημη έγκρισή τους μετά από την ανάγνωση που θα κάνει το Συμβούλιο του σχεδίου προϋπολογισμού που θα γίνει στις 15-16 Ιουλίου. Κλείσαμε με αυτό το σημείο της ημέρησης διάταξης. Περνάμε στο σημείο 15. Θα πρέπει να δώσω το λόγο στην κυρία Ήλντα Φιγιρέντου για την παρουσίαση των τροπολογιών στην έκθεσή της που αφορά που είναι μια έκθεση πρωτοβουλία που αφορά το ρόλο του ελαχίστου εισοδήματο για την κατανόηση τη φτώχεια και την προώθηση μια περιεκτικής και χωρί αποκλεισμού κοινωνία στην Ευρώπη. Έχετε το λόγο, κυρία εισηγήτρια. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, τους και τις συναδέλφους που έχουν παρουσιάσει τροπολογίες στην ε, έκθεση αυτή, καταδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό ότι ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την προβληματική αυτή της ε, επιδίνωσης της ε, ένδυα και του κοινωνικού αποκλεισμού σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και επομένως την εξ αυτής ελκόμενη αναγκαιότητα να προχωρήσουμε προς μια κατεύθυνση η οποία υπερβαίνει τις δηλώσεις καλής θέλησης και καλών προθέσεων μέσα στο έτος αντιμετώπισης της φτώχειας και του αποκλεισμού. Έχουμε λοιπόν ένα πολυπληθές πλήθος τροπολογιών που έχουν κατατεθεί και μέσα από τις οποίες εκφράζονται οι ανησυχίες βουλευτών από διάφορες πολιτικές ομάδες και διάφορους γεωγραφικούς χώρους και εξέρχεται ακόπως η ανάγκη μιας πρότασης μεγαλύτερης σαφήνειας σε ό,τι αφορά το ελάχιστο εισόδημα στα διάφορα κράτη-μέλη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, όπως τονίστηκε και σήμερα το πρωί, είναι απαραίτητη και απαράγραπτη η ανάγκη να κάνω κάποιες εξ αρχής διευκρινήσεις. Αυτό το οποίο επιζητούμε με την έκθεση αυτή πρωτοβουλίας υπογραμμίζω είναι φυσικά το να συμβάλλουμε σε πρακτικό επίπεδο ώστε να επιληθούν τα σοβαρά προβλήματα της ένδυας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δεν μπορούμε να λύσουμε το σύνολο του προβλήματος αυτού. Γνωρίζουμε ότι, όπως λέει και η έκθεση, υπάρχουν διαφορετικές αιτίες για την ένδυα. Πελαμβάνονται στα αίτια αυτά και η κατάσταση των ενδεών εργαζομένων, των οποίων ο αριθμός δεν πάβει να αυξάνεται, όπως ελέγχθηκε προηγουμένως. Και επίσης υπάρχει το πρόβλημα της ανεργίας, του αυξανόμενου αριθμού εργαζομένων που δεν έχουν καμία κοινωνική προστασία, της κατάστασης των ηλικιωμένων πτωχών λόγω των περιορισμένων συντάξεων, των ενδεών λόγω του χαμηλού οικογενειακού εισοδήματο και επομένως έχουμε μια συνολική κατάσταση ένδυας η οποία επιδεινώνεται με την έλλειψη πρόσβασης όχι μονάχα σε εργασία με δικαιώματα αλλά και στις απαραίτητες κοινωνικές υπηρεσίες οι οποίε είναι απαραίτητε σε αυτού που έχουν χαμηλό εισόδημα, όπω είναι η υγειονομική περίθαλψη, η κοινωνική προστασία, η στέγαση, η φτηνή στέγαση, η παιδεία. Είναι λοιπόν αυξανόμενο και ο αριθμό των αστέγων φτωχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτή την έκθεση λοιπόν δεν πρόκειται να δοθεί απάντηση σε όλο αυτό το συνολικό πλέγμα προβλημάτων. Αναφερόμαστε μονάχα στο θέμα της ούτε καν του ελάχιστου μισθού αλλά ενός ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Αυτό καταδεικνύει και τον την περιορισμένη εμβόλια την περιορισμένη εμβέλεια συγγνώμη, αυτής της έκθεσης παρά το γεγονός ότι πραγματεύεται ένα ευρύτατο θέμα. Τονίζεται λοιπόν ότι είναι απαραίτητο μέσα στην δραματική κατάσταση ένδυας ανεξάρτητα από τα αίτια της στην οποία ζουν εκατομμύρια άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μιλάμε τώρα για μια στιγμή που είναι πολύ υψηλή η ανεργία της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντί να είναι η απασχόληση η μόνη απάντηση, δεδομένου ότι υπάρχουν άτομα που δεν μπορούν να εργαστούν, δεδομένου ότι υπάρχουν ηλικιωμένοι, παιδιά, άτομα τα οποία έχουν προβλήματα στον τομέα αυτό, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες αυτές οι συνθήκες και να υπάρξει εγγύηση ενό ελάχιστου εισοδήματο για τα άτομα αυτά που θα του επιτρέψει να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Δεν υποστηρίζω ένα μοναδικό ελάχιστο εισόδημα για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να διαμορφώνεται ανάλογα με τις χώρες. Αλλά διεκδικούμε ένα ελάχιστο εισόδημα το οποίο υπόκειται σε μια κοινή αρχή για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή πρέπει να είναι επαρκέ για να μπορούν τα άτομα να ζήσουν με αξιοπρόπεια και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μέσα στα πλαίσια αυτής της ρύθμιση, της ιδιαιτερότητας όλων των καθεμία από τις χώρες τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν πολλές προτάσεις ειδικά μέσα στι οποίε η ύπαρξη μια οδηγία πλαισίου μέσα από την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να παρουσιάσει προτάσεις οι οποίες θα υπόκειται σε μια σειρά αρχών, μία εκ των οποίων είναι ότι αυτό το ελάχιστο εισόδημα θα μπορούν να είναι το λιγότερο 60% του μέσου εισοδήματος στην χώρα αυτή. Αυτό φυσικά οδηγεί σε ένα διαφορετικό ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά υπάρχει αυτός ο κοινό κόρμος και η κοινή αντιμετώπιση. Αυτό είναι ένα από τα θέματα λοιπόν τα οποία αντιμετωπίζονται σε αυτή την έκθεση. Πρέπει φυσικά να μπούμε σε περισσότερη λεπτομέρεια για ορισμένα από αυτά τα ζητήματα τα οποία περιέχονται σε αυτή την προβληματική και επίσης να δούμε τι γίνεται και με τους στόχους μείωσης της ένδυας. Κάτι την άποψη με αυτό το οποίο κάνει η Κομισιόν σε ό,τι αφορά τη στρατηγική 2020 είναι ανεπαρκές, είναι περιοριστικού χαρακτήρα και δεδομένου ότι μιλάμε για τα επόμενα δέκα χρόνια. Επομένως, <clears throat> πρέπει σε σχέση με αυτή την πρόταση να δούμε ποιες είναι οι δυνατές συμβιβαστικές λύσεις οι οποίες μπορούν να εξευρεθούν με συμφωνία όλων μας γύρω από το θέμα αυτό. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε κοινέ θέσει. Η πλειάδα αυτών των 187 τροπολογιών που διατυπώθηκαν με βρίσκει σύμφωνη, δηλαδή θα υποστηριχθεί από μένα γιατί εξυπηρετούν τον ίδιο το στόχο και ακολουθούν το βασικό πλαίσιο της έκθεσης αυτής. Η συνθλιπτική λοιπόν πλειοψηφία αυτών των τροπολογιών μπορεί να υποστηριχθεί. Απλώς υπάρχουν πολλές επαναλήψεις που υπάρχουν πολλές δηλαδή τροπολογίες που επαναλαμβάνονται μεταξύ τους. Εγώ πιστεύω θα μπορούσα να διατυπώσω τουλάχιστον 12 συμβαστικές τροπολογίες που θα καλύψουν αυτές τις τροπολογίες προσπαθώντας έτσι να, ξαναβρω, να εξεύρω κάποιες λύσεις για την πρώτη παράγραφο όπου υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός τροπολογιών και επίσης σε σχέση με τη δεύτερη παράγραφο που και εκεί υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός τροπολογιών. Σας λέω ότι οι περισσότερες τροπολογίες πηγαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση. Ίσως δεν θα είναι δυνατό να υπάρξει <clears throat> συνένεση όλων γιατί υπάρχουν κάποιε τροπολογίε οι οποίε πηγαίνουν αντίθετα με το ρεύμα. Οι περισσότερε τροπολογίε όμω πηγαίνουν προ μια κοινή κατεύθυνση και υπάρχει δυνατότητα συνένεση και το ίδιο ισχύει και για την παράγραφο 3, όπου και εκεί υπάρχει μεγάλο αριθμό τροπολογιών οι οποίες βρίσκονται σε κοινή κατεύθυνση με μένα. Ακόμα και στην παράγραφο 4 είναι μεγάλος ο αριθμός προτάσεων. Στην 5, 6, 7, επίσης, πιστεύω και στις αιτιολογικές σκέψεις μπορούμε να καταλήξουμε σε τέσσερις προτάσεις συμβιβασμού, μία σε σχέση με την αιτιολογική σκέψη G στα λατινικά, μία σε σχέση με το I το λατινικό, μία σε σχέση με το K λατινικό και μία για το L και μία για το M. Και σε σχέση με αυτά τα οποία περιέχονται στην τωρινή μορφή της εκθέσεως, νομίζω ότι αυτές οι συμβαστικές τροπολογίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για συνένεση μεταξύ των διαφορετικών πολιτικών ομάδων και βουλευτών που κατέθεσαν τροπολογίε. Σα λέω και πάλι ότι υπάρχουν πολλέ νέε τροπολογίε που εισάγουν νέα στοιχεία. κάποιε από αυτέ ακολουθούν την ίδια κατεύθυνση τη έκθεση ή έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα. Εγώ προ το παρόν δεν είχα τη δυνατότητα να δω αν και αυτές θα μπορούσαν να καλυφθούν από συμβαστικές τροπολογίες αλλά έχω μια πρόταση η οποία προήλθε σε, από μια συνάντηση που κάναμε με μερικούς οι οποίοι είχαν καταθέσει τέτοιες τροπολογίες, κάποιοι βουλευτές ή κάποιοι συνεργάτες βουλευτών ήταν παρόντες και θα μπορούσα μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας να σας στείλω ένα πρώτο σχέδιο συμβιβαστικών τροπολογιών, ώστε στις 16 του μηνός στο Στρασβούργο να κάνουμε μια συνεδρίαση η οποία θα εξετάσει αυτό το σχέδιο συμβαστικών τροπολογιών μαζί με τους σχεώδους εισηγητές. Όχι μονάχα σε σχέση και επί τη βάση αυτών των 12 συμβαστικών τροπολογιών στις οποίες αναφέρθηκα, αλλά και για να δούμε κατά πόσο θα μπορούσε να καταστεί δυνατό σε σχέση με τις νέες τροπολογίες, με τις τροπολογίες που συνεισφέρουν νέες προτάσεις για αυτή την έκθεση, αν θα ήταν δυνατόν να υπάρξουν επιπλέον συμβαστικές τροπολογίες για να αποφύγουμε την περιττή επανάληψη προτάσεων οι οποίες είναι μεν εμπλουτιστικού χαρακτήρα για την έκθεση αυτή και μπορούν ως εκ τούτου να γίνουν αποδεκτές και συμφωνώ εξάλλου απόλυτα με αυτές διότι πολλές από αυτές είναι πολύ κοντά στο κείμενο αυτό αλλά είναι απαραίτητο να τις συμπυκνώσουμε σε συμβαστικές λύσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι αν υπάρξουν οι προϋποθέσεις για συμβαστικές λύσεις η ψηφοφορία που θα ακολουθήσει στην Επιτροπή μας τον Ιούνιο θα μπορέσουν να ευδοκιμήσουν και εν πάση περιπτώσει ας αποφασίσει η πλειοψηφία. Αυτά όμως είναι τα θέματα τα κύρια τα οποία νομίζω ότι είναι αυτά για τα οποία μπορούμε να βρούμε κάποια λύση. Ξέρω λοιπόν ότι θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτό το θέμα αυτών των τριών ή τεσσάρων ιδεών που είναι οι βασικές. Το ερώτημα είναι αν πρέπει να υποστηρίξουμε μια οδηγία πλαίσιο που να έχει ένα σύνολο προτάσεων. Υπάρχουν διάφοροι βουλευτές οι οποίοι έχουν υποστηρίξει αυτή την πρόταση και εγώ θα παρουσιάσω μια πρόταση συμβαστική σε σχέση με το θέμα αυτό της ύπαρξης μιας πρότασης για οδηγία πλαίσιο. Το ίδιο ισχύει σε σχέση με τους στόχους μείωσης της ένδυας και το ίδιο ισχύει σε σχέση με τους άλλους τομείς που καλύπτονται προτεραιότητες και πολιτικές που έχουν διατυπωθεί από τις διάφορες πολιτικές ομάδες και σε σχέση επίσης με τα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να πριτανεύουν σε ό,τι αφορά στην ε, παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα αυτά. Εγώ δεν μπορώ να δώσω τώρα λεπτομεριακές ε, απαντήσεις σε καθένα από τους συντάκτες των 187 αυτών τροπολογιών, κάτι το οποίο θα ήταν όπως κατανοείται δύσκολο, αλλά νομίζω ότι καταλάβατε ότι από τη δική μου πλευρά υπάρχει απόλυτο ανοιχτό πνεύμα για να αντιμετωπίσω όλες τις συνεισφορές των συναδέλφων μέσα στο πλαίσιο εφόσον εγγράφονται τις πρότασεις αυτής και φυσικά θα έχω το σκοπό να καλύψω την συντριπτική πλειοψηφία των τροπολογιών οι οποίες θα διατυπωθούν και είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε κυρία Δελίου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρία Φιγκερέντο, με συγχωρείτε που δεν μπόρεσα να παραστώ στη χθεσινή συζήτηση. Υπήρξε μια παρανόηση. Σας συγχαίρω λοιπόν για το έργο σας. Ήθελα οπωσδήποτε να τονίσω διάφορα πράγματα. Πρώτα απ' όλα ότι σήμερα η εργασία και ιδιαίτερα στο εισόδημα από την εργασία δεν προστατεύει από την φτώχεια. Αυτό πρέπει να το θυμίζουμε. Έπειτα, για τη διάρκεια της κρίσης είδαμε ότι τα αυτόματα στοιχεία σταθεροποίησης των ε, δικτύων προστασίας έπαιξαν σημαντικό ρόλο ε, στον περιορισμό των παραγόντων που οδηγούν στη φτώχεια. Όμως αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλά στοιχεία που δεν συγκλίνουν προς αυτό το στόχο στα διάφορα κράτη-μέλη. Έπειτα για την καταπολέμηση και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Ενώ η στρατηγική τη Λισαβόνα ήταν πραγματική αποτυχία, διότι δεν εκριζώσαμε τη φτώχεια και μάλιστα καθόλου, εδώ έχουμε αναλάβει μια ευθύνη ιστορικού χαρακτήρα. Δηλαδή πρέπει εδώ να έχουμε κατά νου και τους στόχους της χιλιετίας του ΟΗΕ. Κυρία Φιγκέρεδο, ξέρω ότι οι πράσινοι θα σας δώσουν πολλή δουλειά να κάνετε. Τις αντικατοπτρίσατε πολλές από τις προτάσεις μας στις συμβαστικές σας αλλά τρει άξονες εδώ μου φαίνονται αποφασιστικής σημασίας για την πορεία που θα ακολουθήσουμε στο μέλλον. Πρώτα απ' όλα ιδιαίτερη μερίμνα για τους νέους, τα πρώτα θύματα της κρίσης αυτούς που είναι συνήθως θύματα της, των διακρίσεων για την πρόσβαση στα κοινωνικά δικαιώματα, όπως στη Γαλλία, τη χώρα μου. Η πρόσβαση στο εισόδημα της ενεργή, ενεργούς αλληλεγγύης έχει να κάνει με το κατόφλι των 25 ετών, για να έχει δηλαδή κανείς δικαίωμα σε αυτό το εισόδημα της ενεργούς αλληλεγγύης. Πρέπει να έχει εργαστεί κανείς δυόμιση χρόνια το λιγότερο και με, υπάρχουν και διάφορες άλλες προποθέσει. Αφορά λοιπόν το 1% των νέων τελικά. Να κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη. <clears throat> Έπειτα πολλές τροπολογίες αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην καταπολέμηση του φαινομένου των αστέγων. Εδώ η έκθεσή σας πρέπει να τονίσει ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η πρόσβαση στις κοινωνικές παροχές για τα άτομα τα οποία είναι τα πλέον περιθωριοποιημένα και τα πλέον ευάλωτα. Να βεβαιωθούμε επίσης ότι ο ορισμός ελάχιστου εισοδήματος ε, λαμβάνει υπόψη το όριο της φτώχειας προκειμένου να εγγυηθεί στον καθέναν επαρκής πόρους για να μπορεί να εξέλθει από τις συνθήκες φτώχειας, να ξεφύγει. Το είπατε κι εσείς, το ελάχιστο εισόδημα πρέπει να είναι ένα δικαίωμα στο οποίο να έχουν πρόσβαση όλοι χωρίς διακρίσεις. Και εδώ έχω υπόψη κατά ιδιαίτερος μάλλον και την κοινότητα των ΡΟΜ. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Δαντέν. Ευχαριστώ. Εκ μέρους της ομάδας μας να σας πω ότι χαιρόμαστε που βλέπουμε ενδιαφέρον από τις διάφορες ομάδες για την έκθεση αυτή. Φαίνεται από τον αριθμό των τροπολογιών. Πολλές ενδιαφέρουσες τροπολογίες, κάτι που περιπλέκει το έργο της εισηγήτριας, όμως αυτές οι ενδιαφέρουσες τροπολογίες πολύ συχνά επικαλύπτονται, αλληλοσυμπληρώνονται. Για παράδειγμα, οι τροπολογίες των πρασίνων της δικής μας ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και της ομάδας ε, Γκουε, της εισηγήτριας δηλαδή. Θα ήθελα λοιπόν να υπογραμμίσω το έργο που έχουμε κάνει. Συναντηθήκαμε χτες και προσπαθήσαμε να βρούμε κάποιους συμβιβασμούς για την συγχώνευση αυτών των ροπολογιών. Το σημαντικό είναι να υπάρξει καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας και αυτό πρέπει να ληφθεί συνολικός υπόψη. Τώρα, για τις τροπολογίες. Καταρχάς, μία ανεκδοτολογική, αν θέλετε, παρένθεση. Ορισμένες φορές είναι προβληματικός ε, προβληματικό το θέμα της μετάφρασης όρων όπως μέσος, ε, μέσος ώρες, ε, moyen, médian στα γαλλικά και δημιουργούνται προβλήματα στην ερμηνεία αυτών των όρων ορισμένες φορές. Η ομάδα μας θεωρεί ότι έχουμε την ευκαιρία να ζητήσουμε μια οδηγία, μια οδηγία πλαίσιο από την Κομισιόν με ένα σύστημα για το ελάχιστο εισόδημα. Δεν χρειάζεται να είναι παντού το ίδιο ελάχιστο εισόδημα, αλλά θέλουμε να έχουμε μια κοινή αναφορά που θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των κρατών μελών. Στα βόρεια κράτη υπήρχε ένα σύστημα με συλλογικές συμβάσεις το οποίο δεν θα έπρεπε να διακινδυνεύσουμε. Αυτό θα έπρεπε να φανεί στην έκθεση. Πέρα όμως από το θέμα της οδηγίας, αυτή η οδηγία για το ελάχιστο εισόδημα που θα έπρεπε να αφορά όλη την Ευρώπη θα έπρεπε να είναι ένα από τα εργαλεία για την καταπολέμηση της φτώχειας και ειδικά των πιο ευάλωτων ομάδων όπως είπε και εκπρόσωπος των Πρασίνων και θα έπρεπε να τονίζουμε την αναγκαιότητα καθολικής πρόσβασης σε ορισμένα βασικά δικαιώματα. Τέλος, να πω ότι ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε σε πνεύμα επικοδομητικό με σας κυρία εισηγήτρια προκειμένου να καταλήξουμε σε έναν καλό συμβιβασμό που θα ανταλαμβάνει όλα αυτά υπόψη του. Η κυρία Λίν, ευχαριστώ. Δεν κατέθεσε τροπολογίες, αν και σκιώδη εισηγήτρια, γιατί μου άρεσε πολύ η αρχική σας έκθεση. Περισσότερο από ότι με τις τροπολογίες. Δεν έχω πρόβλημα με πολλές από τις τροπολογίες, αλλά νομίζω ότι μια πιο επικεντρωμένη και συνοπτική έκθεση είναι καλύτερη. Συμφωνώ με πολλά πράγματα, όμως να πω ότι ορισμένα μέλη της ομάδας μου δεν είναι υπέρ μιας οδηγίας πλαίσιο. Θεωρούν ότι δεν είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Δείτε τι έγινε στην Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία κτλ. Οπότε ίσως δεν θα ήταν καλό να προχωρήσει κάτι τέτοιο τώρα. Άρα παρόλο που πολλοί στηρίζουν την ιδέα αυτή καθ' αυτή, δεν συμφωνούν με την επιλογή της συγκεκριμένης χρονικής στιγμής. Αυτό θα μπορούσαμε να το δούμε για τους συμβιβασμούς. Μετά, το 60%. 60% του μέσου εισοδήματος. Το βλέπω και σκέφτομαι καλή ιδέα. Όμως, σε αυτή την περίπτωση θα αυξηθεί το μέσο εισόδημα, γιατί αυξήθηκε το ελάχιστο εισόδημα, άρα θα πρέπει να αυξηθεί και το ελάχιστο εισόδημα, οπότε πάλι αυξάνεται το μέσο κτλ. κτλ. Άρα θα ήθελα να δω κάτι που θα συσχετίζει το ελάχιστο εισόδημα με το όριο της φτώχειας και να υπάρξει καλός ορισμός του ορίου της φτώχειας. Αντί λοιπόν να μιλήσουμε απλά για 60% του μέσου εισοδήματος. Και θεωρώ ότι η φτώχεια είναι παρόμοια σε πολλά κράτη-μέλη. Αναφέρθηκε στους άστεγους ε, η κυρία Ντελή και εμείς στη χώρα μας προσπαθούμε να θέσουμε στόχους για τη μείωση των αστέγων. Ένας τρόπος είναι το ελάχιστο εισόδημα. Όμως, αν ζητήσετε οδηγία θα χάσετε πολλούς υποστηρικτές που συμφωνούν με τον ελάχιστο εισόδημα αλλά δεν προτιμούν να υπάρξει οδηγία πλαίσιο αυτή τη στιγμή. Εγώ είμαι υπέρ της οδηγίας αλλά θα δημιουργήσει προβλήματα η ομάδα μου και δεν ξέρω αν θα μπορέσει να συμφωνήσει όλη η ομάδα με την οδηγία. Θα μπορούσαμε να το δεχθούμε; αν υπάρξει κάποια διατύπωση που να μιλά για ελάχιστο εισόδημα σε επίπεδο κράτους μέλους, όπως στην αρχική σας έκθεση. Η κυρία Κώστα, παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ιδιαίτερο την κυρία Φιγκερέιδο για το εξαιρετικό της έργο και για την προθυμία να ξεύρει συμβαστικές λύσεις για να γίνει πιο λειτουργικό και το κείμενο και τέλος πάντων να μείνει περιθώριο και για τις τροπολογίες που όλοι θελήσαμε να υποβάλουμε και για να γίνει και πιο ε, καθοριστική στην παρέμβασή της η πρόταση αυτή και πιο αποτελεσματική. Όπως και ο συνάδελφος Κομφεράτη και άλλοι συνάδελφοι υπογράμμισαν, θέλουμε το εργαλείο αυτό να ενδυναμωθεί γιατί έχει και μία συνιστόσα, μία πτυχή πολύ σημαντική κατά της φτώχειας αλλά κυρίως και να αντιμετωπιστεί αυτή η συγκυρία της οικονομικής κρίσης να δοθούν δυνατότητες και θεμέλια για περισσότερη ζήτηση, περισσότερη ανεξαρτησία των πολιτών. Ξέρουμε ότι αυτό που σήμερα λείπει είναι οι επενδύσεις. Χρειάζεται λοιπόν να μειωθεί και η εξάρτηση των ατόμων που έχει και σοβαρό κόστος για τα δημοσιονομικά του κράτους. Η κοινωνική προστασία Άρα χρειάζεται ένα εργαλείο τέτοιο που να χρησιμοποιηθεί ως αθετηρία για να δώσουμε ένα ισχυρό μήνυμα για την αγώνα μας κατά πολέμησης της φτώχειας, αλλά και μέτρα δυνατότητας συμπερίληψης. Καλά είπατε ότι το εργαλείο αυτό θα πρέπει να συμπληρώνει άλλες μορφές υπηρεσιών διευκολύνσεων που θα παρα, παράσχονται ως ένα μείγμα για πιο αποτελεσματική κοινωνική προστασία. Και βάσει της τελευταίας παρέμβασης που άκουσα, πιστεύω ότι η οδηγία πλαίσιο αφήνει στα κρατη και στους κοινωνικούς εταίρους τη δυνατότητα να καθορίσουν και τις πτυχές που σχετίζονται με την ε, πολιτική των επιμέρους κρατομελών. Αυτό δεν έχει μόνο συμβολική αξία, αλλά δίνει και απάντηση σε ένα ζήτημα που μας απασχόλησε πριν από λίγο καιρό. Όταν μιλούσαμε για την ανεργία και την καταπολέμηση της φτώχειας, αλλά δυστυχώς παρέμεινε νεκρό γράμμα ε, ο στόχος αυτός στα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω λοιπόν ότι το εργαλείο αυτό, η όθηση και η ορμή που θα έχουμε μέσα της οδηγίας πλαίσιο, που λαμβάνει βεβαίως υπόψη την επικουρικότητα, θα δώσουμε λοιπόν μια πιο διαρθρωμένη, πιο ανανεωμένη και ίσως και ικανοποιητική απόκριση που θα αφορά και επί επιγενεών πολιτών, πολιτών που έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στα θεσμικά όργανα και θέλουν να δουν την ισχυρή βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναγνωρίσει τα στοιχεία του ανήκειν των πολιτών που έχουν διατυπωθεί και στη συνθήκη της Λισαβόνας. Νομίζω λοιπόν ότι οι τροπολογίες της κυρίας Φιγκέρα εδώ καλύπτουν και αυτή τη συγκεκριμένη περίσταση. Όπως σωστά ανέφεραν και συνάδελφοι από άλλες πολιτικές ομάδες στην Επιτροπή μας. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Βίξον. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μπορώ να πω εξ αρχής ότι εγώ υποστηρίζω κατά 100% τις προσπάθειες μείωσης της ένδυας στην Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι το οποίο φυσικά θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι είναι απαραίτητο. Η Ευρώπη είναι πολυμορφή. Και αναφερθήκαν προηγουμένως στα διαφορετικά συστήματα συλλογικών συμβάσεων. Είναι πολύ σημαντικό όταν έχουμε συστήματα συλλογικών διαπραγματεύσεων και συμβάσεων να το λαμβάνουμε αυτό υπόψη όταν μιλάμε για ελάχιστο ελάχιστες αποδοχές ή ελάχιστο εισόδημα. Μερικές φορές είναι δύσκολο να ξέρουμε ποια είναι η διαφορά μεταξύ των δύο. Ορισμένοι αναφέρονται σε ελάχιστες αποδοχές, άλλοι μιλάνε για ελάχιστο εισόδημα. Πρέπει να είμαστε σαφείς για το πιο ελάχιστο είναι αυτό το οποίο λέμε. Οι ελάχιστες αποδοχές προκύπτουν πολλές φορές από συλλογικές συμβάσεις και αυτό φυσικά είναι ένα σημαντικό εργαλείο και στοιχείο για την καταπολέμηση της ένδυας. Δεν νομίζουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε και δεν θέλουμε να διατρέξουμε τον κίνδυνο να θέσουμε ένα αμφιβόλο της συλλογική και συμβάσει και τι διαπραγματεύσει μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Όπω σα είπα, λοιπόν, είναι μεγάλη ποικιλία στην Ευρώπη και πρέπει να λάβουμε απόψη αυτό το στοιχείο. Ευχαριστώ. Δεν έχω άλλου ομιλητέ εγγεγραμμένου. Θα ξαναδώσω το λίγο, λοιπόν στην κυρία Φιγερέντο για να κλείσει αυτή τη φάση εξέταση εκθέσεώ τη. Εκτός... Ο εκπρόσωπο τη Επιτροπή, θέλετε να σχολιάσετε εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι, η κυρία Φιγκερέιδου λοιπόν. Α, με συγχωρείτε. Μετά, ε, κατόπιν όριμη σκέψεω, η Επιτροπή παίρνει την απόφαση να παρέμβει τελικά. Επιτροπή. Ευχαριστώ. Κάποια γενικά σχόλια, δεν θα απαντήσω σε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Καταρχάς να πούμε ότι η έκθεση όντως ε, δίνει πολιτική όφηση σε αυτό το φάκελο, τον οποίο παρακαλωθούμε στενά. Υπάρχουν κάποια θέματα ε, επί του περιεχομένου, αλλά ίσονος ε, σημασίας, τα οποία οι συνάδελφοί μου θα μπορούσαν να συζητήσουν με τη γραμματεία γραπτός. Δεν θα σας πω τίποτα παρατέρω εδώ. Θα σας στείλουμε κάποια σχόλια επί των περιεχομένων για να σας βοηθήσουμε με την έκθεση. Ευχαριστούμε κυρία Φιγκρέδα για να κλείσουμε. Ευχαριστώ. Απαντώντας στην Επιτροπή, να πω απλώς ότι προτείνω να συμπεριληφθεί μια μικρή αλλαγή ως προς την αιτιολόγηση της συμπερίληψης της σύστασης του 2008. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, όμως αυτό θα παρουσιάζεται και στην έκθεση. Μιλάω για τη σύσταση της Επιτροπής 2008 του, της 3ης Οκτωβρίου. Και αυτό θα γίνει για να καλυφθεί και αυτό το στοιχείο το πιο χειροπιαστό που αναφέρατε. Θα εμφανίζεται στις αιτιολογικές σκέψεις της έκθεσης. Θα υπάρχει αναφορά στο ίδιο το κείμενο, στην αιτιολογική έκθεση. Επίσης να προσθέσω ότι δυστυχώς η σύσταση αυτή δεν είχε τις συνέπειες που επεδίωξε να μας πείσει ότι είχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό έχουμε βρεθεί σήμερα και στη σημερινή κατάσταση. Θα θέλαμε λοιπόν κάτι ισχυρότερο πλέον. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε φτάσει εδώ άλλωστε, για να συζητάμε για ένα πλαίσιο ενίσχυσης των μέτρων αυτών, ώστε να ληφθεί υπόψη η βαρύτητα του προβλήματος ε, του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας σε αυτή τη φάση. Τώρα για τους συναδέλφους που παρενέβησαν και νομίζω ότι από τις τοποθετήσεις όλων έγινε σαφές ότι είναι πολύ δύσκολο και από την πλευρά της κοινοβουλευτικής μας επιτροπής να κατορθώσουμε να πετύχουμε συνένεση για το θέμα μιας οδηγίας, του περιεχομένου της, των στόχων της συνολικά. Ναι, αυτό ισχύει, αλλά θα ήθελα να είναι δυνατό αυτό. Τουλάχιστον αυτό θα επιδιώξω προσωπικά με την εργασία μου και μετά θα δούμε. Και μια σοβαρότατη διευκρίνηση δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή. Επαναλαμβάνω, δεν συζητάμε τώρα για τον ε, ελάχιστο μισθό. Δεν μιλάμε για τις συλλογικές συμβάσεις εδώ. Όχι, σεβόμαστε πλήρως αυτές τις συλλογικές συμβάσεις, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, τον διακανονισμό που ισχύει σε κάθε χώρα. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου συλλογιστική. Ούτε θέλησα να γράψω, ούτε ποτέ να θέσω ένα αμφιβόλο αυτό το σκέλος του θέματος. Έχει να κάνει αυτό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την μεταχείριση της κάθε χώρας για τα μισθολογικά ζητήματα. Αυτό που επιδιώκουμε είναι να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό που να επιτρέπει στα κάτι να εγγυηθούν ένα ελάχιστο εισόδημα. Χωρίς συνεισφορά δηλαδή εισόδημα που δεν θα βασίζεται στην ε, φορολόγηση. Θα προέρχεται όμως από τον προπολογισμό του κάθε κράτους και εδώ η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαγραμματίσει ένα σημαντικό ρόλο μέσω του δικού της του προπολογισμού. ειδικά για τα κράτη που βρίσκονται σε τέτοια δημοσιονομική κατάσταση που μπορεί να χρειάζονται στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που δεν μπορούμε να παραμελούμε είναι το θέμα το σοβαρότατο της φτώχειας, ιδίως της ακραίως, των ακραίων συνθήκων φτώχειας. Θα πρέπει λοιπόν να αναζητήσουμε μια κατάλληλη απόκριση σε αυτό. Επαναλαμβάνω λοιπόν, εδώ δεν μιλάμε για τον ελάχιστο μισθό. Δεν πρόκειται να μπλέξουμε σε αυτή τη διαδικασία. Ούτε τι συλλογικέ συμβάσει θα πειράξουμε, ούτε τι συλλογικέ διαπραγματεύσει καθόλου. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι ένα, είναι ένα ελάχιστο εισόδημα χωρί να υπάρχει συνεισφορά. Και αυτό να προβλέπεται τον προπολογισμό του κάθε εθνικού κράτου. Είτε μέσω του κρατικού προπολογισμού είτε των επιμέρους προπολογισμού αναλόγως με την ιδιαιτερότητα του κάθε κράτους. Και αυτό, επειδή υπάρχουν διαφορετικές ευαισθησίες, τα 70% του μέσου εισοδήματος ε, κατά του 50% του μεσαίου εισοδήματο, αναλόγω με τη διατύπωση που θα επιλέξουμε. Αλλά αυτό το ελάχιστο εισόδημα θα πρέπει να εξασφαλίζει εισόδημα ισοδύναμο με κάτι που να ξεπερνάει το όριο της φτώχειας. Αλλά θα πρέπει εδώ να, ξε... να ξεκαθαρίσουμε και τι εννοούμε με το όριο της φτώχειας. Εγώ προσωπικά αποδέχομαι αυτό που σήμερα ισχύει. Όχι κάτι που κυκλοφορεί και ακούγεται, αυτό που ισχύει σήμερα. Ε, 70% του μέσου εισοδήματος, του μέσου κρατικού εισοδήματος, του κάθε κράτους μέλους, του κάθε εθνικού εισοδήματος. Αυτό λοιπόν μας παραπέμπει σε θέματα ελαχίστων εισοδημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έννοια είναι ελάχιστο εισόδημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλο αυτό. Και στην πράξη θα έχουμε τα ελάχιστο εισοδήματα σε κάθε κράτος μέλος. Αυτά θα διαφέρουν από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Λογικό είναι. Και επίσης πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προϋποθέσεις πρόσβασης στις ε, δημόσιες υπηρεσίες, στις υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας. Υπάρχουν κράτη όπου η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες είναι απλή και άλλα κράτη που είναι σχεδόν αδύνατη η πρόσβαση σε άλλα απολύτως. Πρέπει λοιπόν αυτό να ληφθεί υπόψη. Έτσι, σεβόμενοι τις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας, νομίζω ότι μπορούμε να ορίσουμε ένα πλαίσιο κοινό. Και γι' αυτό ακριβώς αυτό που ήθελα να προτείνω είναι να υποβληθεί επιτέλους αυτή η πρόταση προς την Επιτροπή, να αναλυθεί δράση προς την καταπολέμηση της φτώχεια. Το λέμε πάρα πολύ συχνά στην Ευρώπη. Να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια, το κάνουμε λοιπόν. Σίγουρα πρέπει να γίνει και ανταλλαγή καλών πρακτικών σε πολλά κράτη. Υπάρχουν καλές πρακτικές, σε άλλα πάλι καθόλου. Σε άλλους χρειάζεται στήριξη. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει θέμα για την ελληνική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσω του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Νομίζω ότι αυτό είναι το πλαίσιο εντός του οποίου πρέπει να κινηθούμε. Θα προσπαθήσω λοιπόν να δω και μετά τη συνεδρίαση της 16ης του μήνα με τις νέες προτάσεις και ιδέες που θα ακολουθήσουν θα δούμε τι μπορούμε να καταστρώσουμε. Αυτή είναι η τελική μου τοποθέτηση. Πρόεδρος, ευχαριστώ την εισηγήτρια. Καλό σα κουράγιο για την επεξεργασία των συμβαστικών τροπολογιών. Ψηφοφορία για την έκθεσή σας θα γίνει στις 24 Ιουνίου Έπειτα θα γίνουν διάφορε συνεδριάσει, συναντήσει μάλλον με του ΜΑΝ και του ΔΕ, τους ΔΕ για να επεξεργαστείτε του συμβιβασμού και η έκθεσή σα, όπω θα έχει τροποποιηθεί από την Επιτροπή μα, θα ψηφιστεί τον Οκτώβριο στην Ολομέλεια. Δηλαδή ταυτόχρονα με τη Διεθνή ημέρα, με την Παγκόσμια μάλλον ημέρα κατά τη φτώχεια. Κατά τη διάρκεια τη ημέρα αυτή θα έχουμε και μια επίσημη σύνοδο όπου ο Πολ Μπουσέ έχει προσκληθεί να παρέμβει. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε για σήμερα τη συνεδρίασή μας. Σας ευχαριστώ για την υπομονή, υπομονή σας καθ' τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης. Αύριο η κυρία Λίν ως αντιπρόεδρος θα αναλάβει την πρόεδρια της συνεδρίασης. Καλό σας βράδυ.